Good morning everyone. Καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, μπορούμε να την εγκρίνουμε χωρίς αλλαγές. Μετά έχουμε μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Γεωργίας για τις νέες, τεχνικές, τις νέες ζωοτεχνικές. Στις 17 Μαΐου από τις 10 το πρωί οι νέες ζωοτεχνικές αναφέρονται σε νέες τεχνικές αναπαραγωγής που βασίζονται στις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας και της μοριακής βιολογίας. Μια πολύ αναμενόμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναμένεται τον Μάιο του 2018 για να δούμε κατά πόσον οι ελαιοκράμβοι που είναι ανθεκτικοί στα ε, φυτοφάρμακα μέσω των τεχνικών αυτών μπορεί να περάσει από τη γενική διαδικασία έγκρισης για τα γάματα όμικρον. Ο σκοπός της ακρόασης είναι να δούμε τα θέματα που αφορούν τις νέες τεχνικές ε, αναπαραγωγής και ιδίω τι νομικέ συνέπειε Είναι προσκεκλημένα τα μέλη τη Επιτροπή ΕΕ. Έπειτα, η βιωσιμότητα των συστημάτων υγεία. Σεμινάριο που οργανώνει η Ομάδα εργασία Υγεία. Ε, συμπροεδρεύουν η κυρία Σολεδάτ Καμπεζόν και ο κύριο Ολέης Πέτριλε στι 15 Μαου από τι 10 έω τι 12. Προσκεκλημένα όλα τα μέλη της Επιτροπής ΕΝΒΗ. την 5η 7 Ιουνίου το απόγευμα δεν θα ε, υπάρξει συνεδρίαση, αλλά θα γίνει η πρωινή. Σήμερα έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες και ε, τα κείμενα της συνεδρίασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικώς. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο. Οι συστάσεις των συντονιστών έχουν μοιραστεί ηλεκτρονικώς και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί. Εάν δεν υπάρχουν να τηρήσει στο τέλο της συνεδρίασης, τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη 24 η 25 η ιανουαριου και το 10 η Μαρτίου 2018 θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί και αυτά. Τώρα, στο δεύτερο γύρο ε, τριμερούς διαλόγου για τα ε, λοιπάσματα και το σχετικό κανονισμό στι 11 Απριλίου, την έκθεση Γκαρντίνη, υπήρξαν δύο θέματα επί της ουσίας που συζητήθηκαν, τα όρια του καδμίου και τα παραπροϊόντα. Για το καδμίο, ένα θέμα που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, οι συζητήσεις περιορίστηκαν σε μια παρουσίαση των ε, θέσεων των θεσμικών οργάνων. Σε ό,τι αφορά τα παραπροϊόντα, η συμβαστική πρόταση της Προεδρίας συζητήθηκε και υπήρξε συμφωνία ότι οι περαιτέρω συζητήσεις για την πρόταση αυτή θα ε, διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο. ένας αριθμός τεχνικών αλλαγών στα ε, σχετικά άρθρα συμφωνήθηκαν προσωρινά. Ο επόμενος γύρος του ημερούς διαλόγου έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαΐου. Τώρα, κτηνιατρικά φάρμακα. Η κυρία Γκροστέτ. Ο τέταρτος γύρος ε, ανεπίσημου του ημερούς διαλόγου έλαβε χώρα στις 19 Απριλίου. Σε αυτή τη συζήτηση το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ε, συζήτησαν τα εκκρεμή πολιτικά ζητήματα που αφορούν τις περιβαλλοντικές διατάξεις που ε, εισήχθησαν ως προτάσεις από τις τροπολογίες του κανονισμού. Τα δύο θεσμικά όργανα είχαν εκτενείς συζητήσει για το προσωρινό πακέτο και τη συμφωνία και κοιτάζοντα τι συμβαστικέ λύσει μπορεί να βρεθούν. Ο διάλογο ήταν επικοδομητικό και έγιναν σημαντικέ προσπάθειε και από τι τρει πλευρέ για να ε, συγκλίνουν οι θέσεις και να επιταχθεί συμφωνία. Όμως οι διαπραγματεύσεις ε, δυσκολε... έφτασαν σε δυσκολία διέξοδο σε δύο σημαντικά ζητήματα. Την συμπερίληψη του περιβαλλοντικού κινδύνου και της αξιολόγησής του και τον... για τα προϊόντα που θα εγκριθούν πριν τις 20 Ιουλίου 2000 και τη δυνατότητα του Οργανισμού Φαρμάκων να πιστοποιεί ότι οι παρασκευαστές τρίτων χωρών συμμορφούνται με το ε, δίκαιο της Ένωσης. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφάσισαν να παραπέμψουν τα εκκρεμή ζητήματα για περαιτέρω εξέταση στο τεχνικό επίπεδο με σκοπό να τα επανεξετάσουν στον πέμπτο γύρο τριμερού διαλόγου στις 17 Μαΐου. Τώρα, πρώτο σημείο προσυζήτηση σήμερα το πρωί, ένσταση βάσει του άρθρου 106 για το γενετικο στραποποιημενο ζεχαροτευκλο ζαχαρότευλο H7N. Θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στους συνεισηγητές και μετά σε όσους συναδελφούς θέλουν το λόγο και στην Επιτροπή. Πρώτος μου ομιλητής, ο κύριος Στάς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι και όσοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι εδώ, όντως με διάφορους συναδέλφους από διάφορες πολιτικές ομάδες υποβάλαμε μία ένσταση κατά της ε, ανανέωσης, της έγκρισης ε, για το H7A1, 1 προϊόν ε, το οποίο είναι σαν τη μελάσα, σαν ε, η γρή ζάχαρη, η οποία φτιάχνεται από ζαχαρά το και η οποία χρησιμοποιείται σε ζωτροφές και είναι μία από τις πολλές ενστάσεις που έχουν κατατεθεί. Κύριε Στάσε, μισό λεπτό λέει η Πρόεδρε, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ε, μετάφραση στα αγγλικά, έχει κάποιο πρόβλημα. Αν θα θέλετε παρακαλώ να ελέγξετε κατά πόσο όλα είναι εντάξει. Όλα είναι εντάξει. Κανένα πρόβλημα και αν θα μπορούσατε να ξεκινήσετε. Κανένα πρόβλημα, Πρόεδρε. Συμβαίνουν αυτά. Η ένσταση λοιπόν την οποία υποβάλλουμε μαζί με κάποιους συναδέλφους από διάφορες πολιτικές ομάδες ε, είναι μια ένσταση για την ανανέωση της πιστοποίησης, για την εμπορία, ε, για τρόφιμα και ε, ζωοτροφές του H71, ενώ ζαχαρότευτλο, ένα προϊόν το οποίο είναι σε σιρόπι ζάχαρης, το οποίο παράγεται από ζαχαρότευτλο, αλλά και ε, πολιτό πολτός και μελάς, τα οποία χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές, ε, είναι μία από πολλές ε, ενστάσεις που έχουν κρατεθεί για την εμπορία τέτοιων προϊόντων. Σε διάφορες περιπτώσεις ε, πρόκειται και για ένσταση για την ανανέωση της πιστοποίησης ε, καλλιέργεια τέτοιων προϊόντων. Νομίζω ότι στο ψήφισμα παραθέτονται οι λόγοι για την ένσταση αυτή. Θα το ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα. Ξέρουμε όλοι ότι προκειμένου να δοθεί πιστοποίηση ενός γαμάτα φαόλ μικρών, ε, είτε για να υπάρχει καλλιέργεια, είτε για να καταναλωθεί, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν επιζήμιες ε, συνέπειες και για τον άνθρωπο και για τα ζώα και για το περιβάλλον. Εδώ η ΕΦΣΑ έχει αποφανθεί θετικά σε ό,τι αφορά το προϊόν αυτό και το 2006 όταν ε, δόθηκε η πρώτη πιστοποίηση και το 2017 όταν έγινε έτοιμα για ανανέωση της ε, άδειας αυτής για εμπορία. Αλλά διαπιστώνουμε ότι από τα κράτη-μέλη έρχονται πολλά επικριτικά σχόλια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης σε ό,τι αφορά την ε, ΕΦΣΑ το είχε αγνοήσει και το 2020 και το 2017. Καταρχάς ότι δεν έγιναν δοκιμές σε ό,τι αφορά τις ρίζες και την εισαγωγή αυτών στις ζωοτροφές. Επίσης η μελέτη ε, επίδοση που έγινε επί τρεις εβδομάδες με ε, πρόβατα δεν είναι αντιπροσωπευτική και κάποια κρατημέλη λένε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι η ανθρώπινη έκθεση της πρωτεΐνης ήταν ε, ε, αμεληταία. Επίσης ότι δεν έγιναν δοκιμαστικά πειράματα σε ό,τι αφορά τις αλλεργίες, σε ό,τι αφορά τις ε, μεμονωμένες ε, ότι δεν μας πείθουν τα αποτελέσματα ότι δεν είναι επιζήμιες και ότι επίσης δεν έχουν γίνει αναλύσεις και λείπουν στοιχεία για το φόσφορο και το μαγνήσιο όπως είχε προτείνει όσα. Ξέρουμε λοιπόν ότι αυτό το γάμα το ομικρόν ε, είναι το προϊόν αυτών είναι ατακτικό στη γλυφοσάτη, άρα εκτίθεται σε μεγαλύτερες και επανειλημμένες δόσεις γλυφοσάτης ε, και άρα κατά την ε, συλλογή των προϊόντων αυτών διαπιστώνουμε μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε γλυφοσάτη, το οποίο και μετατρέπει τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Επίσης, οι ρίζες του προϊόντος. Θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον ε, τι γίνεται με τους μεταβολίτες και τις, ε, τα προϊόντα για την καταπολέμηση των ζεζανίων, των ζεζανιοκτώνα. Η ΕΦΣΑ δεν το έλαβε υπόψη αυτό το στοιχείο και όλα αυτά φυσικά εν και τη συζήτηση που έχει γίνει για την γλυφοσάτη. Ξέρω ότι έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση για την γλυφοσάτη, αλλά εν πάση περιπτώσει εστιαστήκαμε σε κακινογόνους ουσίες, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες ε, ε, σκέψεις και φυσικά οι μακροπρόθεσμοι, οι κίνδυνοι στα θηλαστικά, τα προβλήματα που προκαλούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον, η επιρροή στην βιοπικιλότητα και στα οικοσυστήματα. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία προφανώς θα πρέπει να ελεγχθούν και στο άρθρο 4 της ε, οδηγίας για τα βιζονιακτώνα. Και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι μια ανανέωση της εμπορίας ε, του προϊόντος αυτού του Age 71 θα προκαλέσει αύξηση της καλλιέργειας σε άλλες χώρες και νομίζω ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια συγκεκριμένη ευθύνη γιατί είμαστε και ε, μέλη της ε, συνθήκης του ΟΗΕ για τα βιοκτώνα σε ό,τι αφορά την επιρροή στο περιβάλλον. Όταν λοιπόν έχουμε προσπογράψει μια τέτοια συνθήκη και έχουμε δεσμευθεί να μην προκαλούμε ε, ζημιές και προβλήματα στο περιβάλλον, θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί στην πολιτική μας και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα, τα προϊόντα αυτά τα οποία ενδεχομένω μπορεί να προκαλέσουν ε, προβλήματα και στο περιβάλλον και στην υγεία των ζώων και στην υγεία των ανθρώπων. Και τέλος, ε, καταλήγουμε στο ψήφισμα ότι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανταποκριθήκε στα καθήκοντά τη ε, ότι κατέθεσε μια πρόταση η οποία δεν συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ρητάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει αυτή την πρόταση. Ζητούμε εδώ και στην από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει να καταφέρει τα αιτήματα. Μέχρι ότου να προσαρμοστεί η νομοθεσία. Να σας υπενθυμίσω ότι η σε Γιούγκερ το 2014 είχε δηλώσει ότι θα εκδημοκρατήσει τη διαδικασία για την αντιδότηση των γάμματα ομικρών. Ξέρουμε την διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέσει μια πρόταση η οποία ουσιαστικά έβγαλε εκτός ε, παιχνιδιού το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ακόμα ε, κρεμεί. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν καταδεικνύει εκδημοκρατισμό, εκδημοκρατισμό της όλης διαδικασίας και επίσης δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν τηρούνται και οι συμφωνίε για την ιστορική αγορά. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση αυτή την αποσύρει, την οποία την έχει απορρίψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μα καταθέσει μια σοβαρή πρόταση για να ασκήσουμε τα δημοκρατικά μας καθήκοντα, γνωρίζοντας ότι η μόνιμη επιτροπή για τα τρόφιμα εδώ και χρόνια δεν ε, έχει ε, γνωμοδοτήσει, δεν υπάρχει ειδική πλειοψηφία ούτε υπέρ ούτε κατά. Και άρα με όλες τις ενστάσεις που έχουμε καταθέσει και τις οποίες τι τις υποστηρίζει και η Ολομέλεια και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ε, ουσιαστικά επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχει ε, πλειοψηφία δύο τρίτων κατά τη πρόταση. Νομίζω ότι το πολιτικό μήνυμα είναι σαφέ και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα λάβει αυτά υπόψη, να μην συνεχίσει να βασίζεται μόνο σε τυπικά επιχειρήματα και στατιστικέ ε, να καταθέσει στατιστικά στοιχεία για την ε, εμπορία γάμματα ομικρών ε, και να σας πω ότι ε, αυτή η Επιτροπή σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες έχει καταθέσει τρεις φορές πιο πολλές προτάσεις για ανανέωση αδειών γάμματα ομικρών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάνεμπαχ εκ μέρους του κυρίου Μπάλλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να ζητήσω συγγνώμη από τον συνάδελφο Γκουγιον Μπάλλα, ο οποίο δεν μπορούσε να παρευρεθεί σήμερα και θα ήθελα να σα παρουσιάσω την θέση των σοσιαλιστών. Και όλοι μα υποστηρίζουμε αυτά που αναφέρει ο συνάδελφο Μπατιστά. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί και ασέβεια προ το Κοινοβούλιο. Όταν καταντήφονται διαρκώ τέτοιε προτάσει για ανανέωση αδειών, γιατί δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία στον κλάδο αυτό. Στο παρελθόν σε Επιτροπή νομίζω ότι έχουμε παρουσιάσει με σαφήνεια ποιε είναι οι θέσει μας με μεγάλες με μεγάλη πλειοψηφία έχουμε απορρίψει τέτοια αιτήματα για αδειοδοτήσει τέτοιε και η Ολομέλεια και προσπαθούμε να τηρήσουμε τις ε, υποσχέσει που έχουν γίνει και να ακολουθήσουμε δημοκρατικές διαδικασίε, οι οποίες υποστηρίζονται από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου γιατί αυτό δεν ισχύει στην παρούσα φάση σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ. Να έχουμε άλλου συζητητέ. Ο κύριο Χέλνερ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να είμαστε πάλι ευτυχώς Αυτή η παριθμόνα 2455 κάτι τέτοιο ίσως να είναι κάτι που είναι ένα απλά χάσιμο χρόνο. Το ξέρουμε να θα κάνουμε διαδικασία ούτως ή άλλως. Όπως ακούσαμε, αφορά το ζαχαρότεφλο που η το επιστημονικό όργανο που όλοι γνωρίζουμε, είχε εγκρίνει τον Νοέμβριο του 2007 και όπως επίσης όλοι ξέρουμε είχαν πει ότι αυτό το προϊόν είναι ασφαλές όπως και τα αντίστοιχα προϊόντα σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Η Κομισιόν δεν ακύρωσε αυτή την εντολή από ό,τι άκουσα και δεν έχω ακούσει καμία εξήγηση που να με πείθει για την αντίρρηση αυτή. Αντίθετα, η Κομισιόν ακολούσε το πνεύμα της νομοθεσίας, ότι εμεί δηλαδή εδώ θα συναποφασίσουμε με τις χώρες μέλη. Και χαίρομαι που είχε εγκριθεί στο Συμβούλιο αυτή η νομοθεσία όταν είχαμε τους περισσότερους πράσινους υπουργούς στην ιστορία που έκαναν ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνουν λόγω νομοθεσίας αλλά τελικά φαίνεται δεν έχει σημασία τι λέει η ΕΦΣΑ ή το Συμβούλιο, επειδή εδώ υπάρχει στην Επιτροπή μας πλειοψηφία, η οποία δεν επιθυμεί τη διάθεση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων στην αγορά. Και αυτό οδήγησε σε αυτές τις ε, αναλυθείς, στους αναλυθείς ισχυρισμούς για αυτό το συμβουλιο επειδη εδω υπαρχει στην επιτροπη μας πλειοψηφια η οποια δεν επιθυμει τη διαθεση γενικά ανθρωποποιημενων προιοντων κατά την απόψή μου. για την γλυφοζάτη. Θεωρώ το συγκεκριμένο είναι ανθεκτικό στην γλυφοζάτη. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποια ίχνη γλυφοσάτη, αλλά έχουμε κάποια όρια. Ξέρω ότι έχουμε μια μεγάλη συζήτηση για τη γλυφοσάτη, αλλά α μην μετατρέψουμε σε συζήτηση για τη γλυφοσάτη. Γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι νόμιμη η γλυφοσάτη. Και Όπω ξέρετε, θέλω έτσι να είμαι κάπω προκλητικό και θα είμαι προκλητικό σε αυτή την περίπτωση. Εδώ υπάρχει μια απεικιοκρατική αιτίαση που λέει ότι τέλος πάντων εμείς για τα παραπροϊόντα έχουμε ευθύνες. Ναι βεβαίως έχουμε ευθύνες σε σχέση με τις τρίτες χώρες, όμως πιστεύω δεν έχουμε δικαίωμα να νομοθετήσουμε για το πώς ακριβώς αυτά θα παράγονται στις τρίτες χώρες. Αν αυτές δεν θέλουν να το παράξουν, θα το παράξουν άσχετα αν θέλουμε εμείς να το καταναλώσουμε ή όχι. Αλλά ο ισχυρισμό εδώ πέρα που συνοδεύει αυτή την αντίρρηση δεν βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνουμε ακριβώ το αντίθετο. Το τελείω αντίθετο από αυτό που λέει και τεκμηριώνει ή ισχυρίζεται η αντίρρηση. Θα πρέπει να κάνει εύσα ό,τι πρέπει, το ίδιο και η Κομισιόν και έτσι θα αποδεχτούμε την πρόταση. Το Συμβούλιο, δεν ξέρω κατά πώ το Συμβούλιο κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει. Πάντω είναι ενδιαφέρον ότι η αναφορά στο Συμβούλιο, σε αυτή την αντίρρηση, διαφέρει από τις υπόλοιπε που έχουμε συνήθω. Λέει τέλο πάντων το Συμβούλιο δεν γνωμοδότησε, το οποίο εντάξει ισχύει σήμερα, αλλά συνήθω αναφέρονται και τα αποτέλεσματα τη ψηφοφορία. Εδώ θα θέλω να μάθω γιατί δεν αναφέρονται, δεν παρατίθενται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο, σε αυτή την αντίρρηση. 0,41% απόσταση δηλαδή σε ψήφους ή έλειπαν ψήφοι σε σχέση με την ειδική πλειοψηφία όταν υπερψήφισαν για χώρες κλπ. Εγώ θα έλεγα λοιπόν σήμερα ότι είναι σημαντικό τρόπο ποτέ να έχουμε επιστημονικές αποδείξεις για τη χρήση αυτών των προϊόντων, αλλά να μην πηγαίνουμε παραπέρα. Και όταν λέω ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε σε επιστημονικά τεκμήρια, εννοώ προερχόμενα από τους αρμόδιους επιστημονικούς οργανισμούς. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν διαφορές μεταξύ επιστημόνων Οπότε θεωρώ λοιπόν ότι το λογικό για μας ως σώμα θα ήταν να απορρίψουμε αυτή την αντίρρηση για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ κύριε Μιλιό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτά που είπαν οι προλύσαντες ε, με παρότριναν να ε, συμμετάσχω και εγώ στη συζήτηση. Πρώτα το γεγονός ότι η κυρία Κάντιμπαχ και ο κύριος Στάς ε, παρουσίασαν όλα τα επιχειρήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε και σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματα των πρασίνων και των σοσιαλιστών. Δύο στοιχεία θα ήθελα να κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά. Έχουμε τα στοιχεία για την γλυφοσάτη και είπατε ε, τι έκανε η ΕΦΣΑ, ποια ήταν τα επιστημονικά πορίσματα. Δεν θα ήθελα καν να επισέλθω στα στοιχεία αυτά. Η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια αυτών των ζαχαροτευτλών. Και έτσι λοιπόν επιμολύνεται τα χωράφια. Όταν λοιπόν χρησιμοποιείτε τέτοια γλυφοσάτη, να είστε σίγουροι ότι ε, αν χρησιμοποιείτε εκεί γλυφοσάτη, χρησιμοποιείτε και αλλού γλυφοσάτη. Όλη αυτή η συζήτηση για τη γλυφοσάτη στη Γερμανία αναφέρεται και στην ε, προετοιμασία του εδάφους με τα Όταν όμως ε, γίνεται κάτι τέτοιο, είναι σαφές ότι συνεχίζεται η χρήση της γλυφοσάτης και στη συνέχεια. Και όλοι γνωρίζουμε ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα της ΕΦΣΑ, αυτό έχει σημαντικές ε, επιπτώσεις στην βιοπικιλότητα. Ούτε εσείς δεν θα μπορέσετε να καταπολεμήσετε αυτό ως θεωρία, γιατί υπάρχουν σαφή αποστημονικά απορίσματα που έχουν παρουσιαστεί σε πολλές επιτροπές. Αν λοιπόν κάτι θέλουμε να κάνουμε και να το καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα διδανειοκτώνα και πώς τα χρησιμοποιούμε. Και κάτι άλλο. Γίνεται διαρκώς αυτό το παιχνίδι πινκ-πονγκ. Και εδώ κοιτώ προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θέλουμε σαφήνεια. Σε ό,τι αφορά τον τύπη ζημούν τα κράτη-μέλη. Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουμε σε επίπεδο επιτροπή. Και αυτό το σημείο κριτική θα ήθελα να το έχω αναφέρει. Ευχαριστώ. Άλλο κανεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι από την αρχή της θητείας μου στην Επιτροπή έβλεπα ότι είχαμε δύο διλήμματα. γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και παρουσία τους στα τρόφιμα μας, κάτι το οποίο ήταν ανέκαθεν προβληματικό και δεν υπάρχει διχασμός γιατί περισσότεροι είμαστε κατά. Με κάποιες εξαιρέσεις τέλο πάντων. Και άλλο ένα ζήτημα το οποίο επανέρχεται τακτικά είναι η γλυφοσάτη. Η κατάσταση έχει ως εξής. Έχουμε μια μεγάλη πολυεθνική που ασχολείται με την βιοτεχνολογία και παράγει ένα πολύ ισχυρό ζυζανιοκτόνο το οποίο είναι αποτελεσματικό για πολλά φυτά και μετά έχουμε και το θέμα των γενικά τροποποιημένων προϊόντων όπως η σόγια ή όπως αυτό εδώ το ζαχαρότεφλο, όπου η αποτελεσματικότητα αυτού του προϊόντος είναι μικρότερη. Η γλυφοσάτη λοιπόν όντω είναι κάτι το προβληματικό επειδή προκαλεί καρκίνο, παραμένει στο έδαφος, παρόλο που αυτό το συγκεκριμένο σημείο δεν συνοδεύεται από απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι παραμείνει στις ρίζες των φυτών. Αλλά τέλο πάντων, νομίζω ότι ανεξάρτητα με το τι θα αποφασίσουμε εμείς να κάνουμε εδώ, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των συστημάτων μας. Ευτυχώ τώρα έχουμε μια ειδική επιτροπή η οποία θα εξετάσει την αδειοδότηση για κάποια ζυζανιοκτώνα. Η επιτροπή η οποία έχει συγκροθεί από την Επιτροπή θα περιμένουμε όμως, θα περιμένουμε όμως ένα οχτάμινο μέχρι να λάβουμε την τελική τους έκθεση. Προς το παρόν λοιπόν εμείς ως ομάδα ECR αποφασίσαμε να υπερψηφίσουμε την πρόταση αυτή για την υιοθέτηση αυτή τη αντίρρησης γιατί παραμένουν ακόμα πολλά ερωτηματικά όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και θεωρώ ότι και τα θέματα δημόσιας υγείας έχουν τεράστια σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πίρικ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, δεν σκοπεύω να πάρω το λόγο. Αλλά παρ' όλα αυτά θέλω να πω το εξή. Εδώ και χρόνια το συζητάμε το θέμα αυτό. Η ΕΦΣΑ συμφωνεί, η Επιτροπή συμφωνεί. Και αυτό που είναι σαφέ είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει και παραγωγή τροφίμων. Πρέπει να συμβεί και αυτό. Ωραία και καλά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ο, ο άνθρωπο πρέπει να φάει. Και ο αγρότη κάνει όλο και πιο πολύ ότι μπορεί για να βρίσκει τις καλύτερες πρακτικές για να παράγει τρόφιμα και χρειάζεται σαφήνεια. Ως τώρα, εγώ λοιπόν την, ε, τα επιστημονικά ιδρύματα υποστηρίζω και ρωτώ λοιπόν το εξή συγκεκριμένο. Και οι επιχειρηματίες έχουν θέσει λοιπόν αυτό το θέμα, αλλά και άλλα. Όλοι αναζητούμε πράσινα ε, προϊόντα τα οποία δεν παίρνουν ε, αντιοδότηση. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτή η παραγωγή τροφίμων. Εγώ λοιπόν υποστηρίζω αυτά που λέει ο κύριος Φιέλνερ, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι η συνέχεια που θα δοθεί στο θέμα αυτό, γιατί ο κόσμος το θέτευε το ερώτημα. Uh, Ευχαριστούμε. Και τώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, κύριε και κύριοι βουλευτές, για τα σχόλιά σας. Για άλλη μια φορά, με μεγάλη προσοχή και σεβασμό, ακούσαμε όλες αυτά τα σχόλια, παρόλο που είμαστε στο πλαίσιο της, ε, του ελέγχου και της παρακολούθησης της όλης διαδικασίας, το περιεχόμενο της συζήτησης. Προϊόν από γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότατο. Δεν υπάρχουν ε, ζώντα, ζώντες γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί. Έχει επιτραπεί για σκοπούς σύντησης και για ζωοτροφές. Είναι ήδη παρασκευασμένο όταν το εισάγουμε, οπότε μπορούν και οι γεωργοί και οι καταναλωτές είτε να αγοράσουν το προϊόν είτε όχι, διότι υπάρχει σχετική επισήμανση σε ορισμένους τομείς κάποιοι γεωργοί ε, εισάγουν το προϊόν αυτό διότι μάλλον το χρειάζονται κάπου. Άρα οπωσδήποτε μπορεί η αγορά η ίδια, ο οικονομικός κλάδος, να αποφασίσει αν θα πετάξει αυτό το προϊόν ή όχι αλλά προφανώς κάποιοι το θεωρούν χρήσιμο. Ο ρόλος των αρμόδιων αρχών είναι να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα αυτά, εφόσον εισάγονται, είναι ασφαλή. Γι' αυτό έχουμε αυτό το σύστημα παρακολούθησης. Σε ό,τι αφορά την γλυφοσάτη, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συζητήσεις, το μέγιστο όριο για κατάλοιπα έχει οριστεί για όλα τα προϊόντα. Είτε είναι προϊόντα που παρασκευάζονται εντό Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εκτό. Αυτό το μέγιστο επίπεδο καταλήπων, το MRL, υπάρχει και για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού. Οπότε, όταν εισάγονται τέτοια προϊόντα, πρέπει να έχουν τη σχετική επισήμανση, και να σέβονται το μέγιστο ο επιτρεπόμενο όριο. Κάτι που δεν ορίζεται στον κανονισμό για τα γάματα φόμικρα, γάματα φόμικρα αλλά στα φυτοφάρμακα και στους ζανιοκτώνα και το σχετικό κανονισμό για σκοπούς συνοχής. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει θέμα για την ασφάλεια των ε, τροφίμων και ζωοτροφών. Εμείς το ε, ρυθμίζουμε και οι καταναλωτές έχουν και την επιλογή εάν θα αγοράσουν το προϊόν ή όχι. Την επισήμανση την έχουν. Το ίδιο και για την κοινότητα των γεωργών και κτηνοτρόφων. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, μπορώ απλώς να πω ξανά και εκ νέου ότι έχουμε ακολουθήσει όλα τα βήματα της διαδικασίας. Η ΕΦΣΑ έχει εκπονήσει σχετική αξιολόγηση κινδύνου και δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος που να έχει εντοπιστεί. Επίσης δημόσιες διαβουλεύσεις έγιναν και η ΕΦΣΑ σχολίασε όλες τις απόψεις των δημοσίων διαβουλεύσεων και οι σχετικές πληροφορίες έχουν δημοσιοποιηθεί. Οι διαβουλεύσεις βεβαίως έγινε με συμμετέχοντες από τα κράτη-μέλη και το ευρύτερο κοινό. Όπως ήδη υπόθηκε από κάποιους από εσά, η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στην Επιτροπή, δεν, υπάρξει, υπήρξε καμία γνωμοδότηση, παρόλο που ήμασταν στα όρια της ενισχυμένη πλειοψηφία. και βάσει της διαδικασίας TEPS η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ακολουθήσει τους κανόνες της επιτροπολογία και να υποβάλει πρόταση στην Επιτροπή Ένη. στην Επιτροπή Εφέσεων. Η Επιτροπή αυτή που εξετάζει τις εφέσεις ε, συνέρχεται σήμερα. Ως προς τα ζητήματα της βιοποικιλότητας πρέπει να βεβαιωθούμε ότι, να παραδεχτούμε μάλλον ότι οι τρίτες χώρες είναι και αυτές ε, κυρίαρχες, εθνικώς κυρίαρχες και είναι και συμβαλόμενα μέρη στη σύμβαση της βιοποικιλότητας δεν θα πρέπει να βρίσκουμε πρόσχημα τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς για να καταγγείλουμε τρίτες χώρες ότι δεν σέβονται τη φύση. Υπάρχουν υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και άλλες συμφωνίες, οπότε δεν μπορούμε με την αφορμή της εξουσιοδότησης ενός προϊόντος που έχει ακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα βήματα της διαδικασίας να κουνάμε το δάχτυλο σε τρίτες χώρες και να τους λέμε ότι πρέπει να κάνουν κάτι άλλο από αυτό που κάνουν. Έχω ακούσει και τα περί δημοκρατικού ελλείμματος που κάποιοι από εσάς υπογραμμίσατε, αλλά πολλά κράτη-μέλη είτε καταψηφίζουν είτε απέχουν. Παρόλο που η κοινότητα των γεωργών και κτηνοτρόφων σε αυτά τα κράτη-μέλη εισάγει το εν λόγω προϊόν. Εκεί βλέπουμε το δημοκρατικό έλλειμμα, διότι θεωρούμε ότι στα κράτη-μέλη που υπάρχει καταψήφιση ή αποχή, το πρόβλημα είναι σε εθνικό επίπεδο. Η δυνατότητα λοιπόν που έχουμε δώσει στα κράτη-μέλη στην πρότασή μας να ε, αποφύγουν την εισαγωγή αυτών των προϊόντων θα έπρεπε να αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την άποψή μας είναι απάντηση στο δημοκρατικό έλλειμμα τουλάχιστον όπως το εκλαμβάνουν κάποιοι πολίτες. Την πρόταση αυτή δεν την απέρριψε το Συμβούλιο, ακόμη συζητιέται στις σχετικές ομάδες εργασίας, έχει απορριφθεί όμως δυστυχώς από αυτό το σώμα. Σε ό,τι αφορά την έκκληση να μην εγκριθούν άλλοι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί μέχρι τη διαδικασία της επιτροπολογίας, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσουμε αυτή την ε, προτροπή. Διότι αυτό σημαίνει ότι μόλις κάνει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τροποποίηση σε υπάρχον νομοθέτημα, το υπάρχον νομοθέτημα δεν θα ισχύει πλέον. Αυτό θα έδινε μια ε, εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στην ουσία θα έπρεπε να βρίσκεται στα χέρια του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Άρα, προφανώ μέχρι να εγκριθεί πλήρω από αυτό το Σώμα και το Συμβούλιο η πρόταση αυτή, θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Ε, εν είδη συμπεράσματο, λοιπόν, δεν μπορούμε να δεχτούμε να αποσύρουμε αυτό το σχέδιο απόφαση βάσει και τη νομοδότηση τη ΕΦΣΑ και των κανόνων της ε, διαδικασίας. Και θα επαναλάβω και πάλι εν είδη συμπεράσματος ότι δεν μπορούμε να ε, υπερβούμε τις υποχρεώσεις εφαρμογής της νομοθεσίας. Ευχαρίστως φυσικά να ερχόμαστε εδώ και να συζητάμε τις απόψεις σας, όμως θα καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ακολουθήσαμε όση επιτάσσει η νομοθεσία, είμαστε πλήρως ομορφούμενοι με το περιεχόμενο και τα διαδικαστικά βήματα που αναμένεται να ακολουθήσουμε. Και ελπίζω ότι με τις εξηγήσεις αυτές που μόλις σας δόθηκαν έχω καλύψει τις ε, ανησυχίες σας. Ελπίζω τουλάχιστον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας στο ζήτημα αυτό. Θα ψηφίσουμε το ή άλλο σήμερα το απόγευμα επί του θέματος. Επόμενο. Ένταση. Και πάλι βάση του άρθρου 106. Έγκριση για μέγιστα επίπεδα καταλήπων MRL για τις εξής ε, ουσίες. Τις βλέπετε στον τίτλο, δεν θα μπω καν στην προσπάθεια για ε, την περιεκτικότητα ε, σε κάποια προϊόντα. Σχέδιο ψηφίσματος ακολουθεί και η εισηγήτρια ε, είναι η κυρία Γκοντά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου που επέτρεψαν να συνταχθεί γρήγορα η ένσταση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ προτείνει να αυξηθούν τα ανώτατα όρια 17 ενεργών ουσιών σε γεωργικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το σουλφοξαφλόρ. Προτείνει το ανώτατο όριο να επιτραπεί ε, στα αμπέλια 200 φορές και στις αγκινάρες επίσης να αυξηθεί πάρα πολύ. Το 2015 είχαμε υποβάλει ένσταση για την έγκριση του σουλφοξαφλόρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή ήταν μια νέα κατηγορία νέων νοικοτινοειδούς και ε, μάλιστα πρώτης γενιάς. Αυτό πλήττει το κεντρικό νευρικό σύστημα των μελισσών. Εκείνη την εποχή δεν είχε γίνει δεκτή η ένσταση, απερίφθη με 31 ψήφους κατά, 18 υπέρ, και μία εποχή για λόγους ε, που ήταν ε, πολιτικοί και αρκετά ε, καταδικαστέοι, εφόσον έχουν να κάνουν με το κόμμα από το οποίο προέρχομαι, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη υγεία των μέλισσών και υπεραιτέρω περαιτέρω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα ακολουθήσαμε τις σχετικέ πολιτικές και διαδικαστικές διαδικασίε. το Νοέμβριο στη Γαλλία, το Διοικητικό Δικαστήριο τη Νίκαια ακολούθησε την πρότασή μου για ασφαλιστικά μέτρα και ζήτησε την αναστολή της χρήσης δύο ε, ε, ζυζανιοκτώνων. Ε, το δικαστήριο θεώρησε ότι ήταν άμεσος ο κίνδυνος για την δημόσια υγεία και τις μέλησες. Πριν από τέσσερις μέρες, στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση, πέρασε μία τροπολογία ζητώντας να επεκταθεί το πεδίο των νοικοτινοειδών, περιλαμβάνοντας χημικές ουσίες, ακόμη και αν δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί ως τέτοιες, και να θεωρηθούν ακριβώς νέο νοικοτινοειδή όπως το σουλφοξαφλόρ. Υπάρχει λοιπόν κινητοποίηση και από την πλευρά της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτικών για να καταγγείλουν τον κίνδυνο που αποτελεί το προϊόν αυτό για τις μέλισσες. Η Επιτροπή μας δεν μπορεί να ε, μην ακολουθήσει αυτή την τάση και δεν μπορούμε να δεχτούμε την αύξηση των αντατών ορίων στο Ξαφλόρ, στα αμπέλια και τις αγκινάρες θα πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να ε, λάβει γνώση του φαινομένου της ε, φθήνουσας τάσης του πληθυσμού των επιπολαστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή των μελισσών. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι εναλλακτικέ μπορούμε να έχουμε για το λίπασμα αυτό, για το φυτοφάρμακο αυτό, και να είναι πιο παραδεκτέ. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τον πληθυσμό των μελισσών διαρκώ να μειώνεται. Είναι απαράδεκτο. Οι μέλισσε είναι απαραίτητες για τη διατήρηση του οικοσυστήματό μα. Αν ε, ε ξαλειφθούν θα υπάρξουν βαρύτατε συνέπειε για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ζητώ συνάδελφοι να στηρίξετε για τις μέλισσε και την υγεία μα αυτήν την έκταση. Σα ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. See κάποιος άλλος για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι ο κύριος Φέλτερ. Πια θα μιλήσω ως Judy Gerling την οποία αντικαθιστώ βεβαίω ή εκπροσωπώ. θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Η κυρία Gerling λοιπόν, και εγώ ίδιος βεβαίω, και το αλκοολόκληρο, προτείνουμε να μην στηρίξουμε αυτή την ε, πρόταση ψηφίσματος και θα σας παραθέσω την επιχειρηματολογία. Καταρχάς έχουμε την Επιτροπή, την αρμόδια, η οποία έδωσε τη σύμφωνη γνώμη προς την Επιτροπή για την μείωση των ορίων. Η ΕΦΣΑ επίσης πρότεινε αυτά τα ανώτατα όρια σε σχέση βέβαια με την υγεία των καταναλωτών. Επιπλέον, αυτό η πρόταση ψηφίσματος παραθέτει αναλυθεί στοιχεία σε σχέση με τις ουσίες αυτές και κυρίως του σουλφοξαφλόρ. Στην, ε, στην παράγραφο αναφέρει σωστά ο συντάκτης ότι αυτή η ουσία σουλφοξαφλόρ ανήκει σε αυτή την γενικότερη τάξη των ε, σουλφοξαφλοειδών, όμως δεν ανήκει στα νοικοτινοειδή λόγω ακριβώς τη χημικής σύστασης και είναι, ανήκει σε διαφορετική χημική κατηγορία. Και μάλιστα στην C αναφέρεται ότι η ΕΦΣΑ δεν έχει ταξινομήσει, δεν έχει κατατάξει το σουλφοξαφό ως νοικοτινοειδέ. και ως εκ Είναι δασμένες οι παραπομπές του Σιντάκη ότι τα νεονικοτινοειδή είναι βλαβερά. Παράξενα λέω το γεγονός ότι η ΕΦΣΑ δεν έχει ταξινομήσει, δεν έχει κατατάξει το ασούλφοξαλφόστανε στα νοικοτινοειδή. Επίσης έχουμε και την απόφαση ενός δικαστηρίου στην Ίκαια. Εντάξει, μπορεί να μας αρέσει. Και έχουμε και μια πρόταση από την Κομισιόν για τα ανώτατα επιτρεπτά όρια τα οποία καθορίζονται όταν έχουμε επιπτώσεις στην υγεία των ανθρωπίνων όντων και όταν έχουμε παράγωγα προϊόντα όπως το μέλι. Οι αλλαγέ λοιπόν στα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτή την περίπτωση, δεν θα έχουν επιπτώσεις στην υγεία των μελισσών. Γιατί εμείς συνήθω νομοθετούμε και θέτουμε μέγιστα επιτρεπτά όρια για την υγεία των ανθρώπων. Είναι τελείως διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο ό,τι αφορά της μεση 1107 1107-2009 όσον αφορά διάθεση στο εμπόριο φυτικών ή άλλων προϊόντων. Επιπλέον, το σουλφοξαφλόρ είναι νέο προϊόν, οπότε κατά συνέπεια δεν είναι απαραίτητο η αλλων προιοντων επιπλεον το σουφοξαφλορ ειναι νεο όπως η γεωργική βιομηχανία, να το ρυθμίσει από τώρα. Επίσης, οι παραπομπές στην παράγραφο 5 για τα νεονικοτινοειδή ω ομοιογενής ομάδα, τα οποία θα πρέπει ομού να εγκριθούν ή να απορριφθούν. Εμείς προτιμούμε αντίθετα το τωρινό σύστημα όπου οι ουσίες εξετάζονται κατά περίπτωση, οπότε η παράγραφος 5 δεν είναι σωστή. Να πω και για το προσωπικό. Αυτό ακολουθεί και ένα σχήμα που δείχνει ότι συνήθως έχουμε δύο επιτροπές που αξιολογούν αυτές τις ουσίες και στην ουσία ακυρώνουμε τη δουλειά τους αν δεχτούμε αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Αν αυτό κάνουμε για τα σοβαρά, τα δύσκολα ζητήματα, τότε καλύτερα να τις καταργήσουμε αυτές τις μόνιμες επιτροπές και να περνάμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες, χωρίς καμία τεχνογνωσία ή συμβουλή. Γιατί φαίνεται ότι αυτές οι επιστημονικές ενδείξει δεν έχουν και τόσο νόημα. Δεν νοιάζουν και τόσο κάποια μέλη εδώ πέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε και ο Σπόρος. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Για τις ουσίες που συζητάμε. και το σουλφοξαφλό συγκεκριμένα τέθηκε σε ισχύ πριν τρία χρόνια. Η ΕΦΣΑ κατέληξε ότι τα διαθέσιμα δεδομένα ήταν ανεπαρκή για να αποκλείσουν υψηλό κίνδυνο σε σχέση με το μέλι και τις μέλισσες. Βλέπαμε λοιπόν ότι εγκρίθηκε το σλοφοξαφλόρ παρά τις εκτιμήσεις για τον κίνδυνο. Και η Κομισιόν και η Αρμόδια Επιτροπή είπαν δεν είχαν επαρκή στοιχεία, όλα αυτά έδωσαν έγκριση. Και αυτό είναι σε αντίθεση με την αρχή της απαγορεύσης των ζυζανιοκτώνων ε, για τα οποία λέμε ότι όταν έχουμε παρόμοια δράση όπως τα νεονικοτινοειδή λόγω ακριβώς του κινδύνου στις μέλισσες και το μέλι. Η έγκριση λοιπόν του Ουλσού Foxanflor είναι επίμαχη, αλλά κατέληξε η ΕΦΣΑ λέγοντας ότι έχουμε κατάλοιπα του σουλφοξαφλόρ στα Μπελόφυλλα και σε άλλα φυτά. Οπότε Δεν μπορούμε νομίζω να ανατρέψουμε την απόφαση του 2015 λόγω ακριβώ αυτή τη απόφαση τη ΕΦΣΑ. Γιατί το, η συγκεκριμένη ουσία είναι εγκεκριμένη. Τώρα, τούτου λεχθέντο, έχω και μία ερώτηση προ την Επιτροπή. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγηση από το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας, η έγκριση του σουλφοξαφλόρ δεν περιορίζεται, περιορίζεται σε συγκεκριμένε χρήσει. Θα έπρεπε να είχε να είχαν υποβληθεί επιπλέον στοιχεία που αφορούν ακριβώς τις μέλισσες και την έκθεση όσον αφορά την, επικονίαση. Πρέπει λοιπόν να δούμε εδώ τι γίνεται με τους κινδύνους, τους επικονιαστές, εκτός μελισσών. Οι χώρες μέλη και η αρμόδια αρχή ε, είχε προθεσμία, είχαν προθεσμία μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Μπορεί λοιπόν η Κομισιόν να μας ενημερώσει σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ κύριε Ριβαζή τώρα. Merci, Madame la Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτές οι ενεργές ουσίες και συγκεκριμένα το σουλφοξαφλόρ είναι ενεργέ ουσίες παρόλο που δεν έχουν ταξινομηθεί ως νεονικοτινοειδή. Όπως είπε ο συναδελφό, έχουν τον ίδιο τρόπο δράση. Και στη Γαλλία όπως είπαμε στις 20 Απρίλη είχα μια τροπολογία που έλεγε ότι θα πρέπει να θεωρηθεί νεονικοτινοειδέ. επειδή έχει ακριβώς την ίδια δράση. Δηλαδή στου λήπτε του νευρικού συστήματο των εντόμων. Οπότε ε, δρά ως ε, ως παρασιτοκτόνο. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται τώρα με το επίπεδο των καταλήπων. Έχουμε το κείμενο της απόφασης του δικαστηρίου, γιατί όπως είπαμε ήταν δικαστηρίο στην Νίκη της Γαλλίας, που αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις σε σχέση με τη χρήση. Αναφέρει ότι η έγκριση για διάθεση στην αγορά αυτού του προϊόντος που δόθηκε στην επιχείρηση DAO SAS δεν διασφαλίζει με ασφάλεια ούτε τη συμμόρφωση όσον αφορά τις εμπορικές ε, ε, και επαγγελματικέ προδιαγραφές, ούτε σωστή χρήση αυτού του προϊόντος, ούτε την ε, διασφάλιση του ότι η χρήση η οποία χρησιμοποιείται δεν αποτελεί κίνδυνο για τις μέλησες και για τη δημόσια υγεία. Το είπε λοιπόν αυτό το δικαστήριο, οπότε σύμφωνα με ένα αρχή λοιπόν αυτή της ε, επιφύλαξης που βρίσκεται και στην Συνθήκη Ευρωπαϊκή και στο Γαλλικό το Σύνταγμα, σταματήσαμε αυτή την διάθεση. Αυτή λοιπόν η ενεργό ουσία έχει σταματήσει να διατίθεται στην Γαλλία, επειδή ακριβώ έχει επιρροές στι μέλισσε. Έχει λοιπόν τον ίδιο τρόπο δράσης, ενώ εμείς την εγκρίνουμε, την εγκρίνουμε το 2015 τη στιγμή που έχει αποφασίσει το Γαλλικό Δικαστήριο να την απαγορεύσει. Είναι ένα προϊόν λοιπόν το οποίο να σα πω επίση ότι είναι απαγορευμένο στη ΣΥΠΑ. Ενώ εμεί εδώ στην Ευρώπη θέλουμε να προστατεύσουμε περισσότερο, οι Αμερικανοί το απαγορεύουν. Πώ θα, κάνουμε, λοιπόν, θα προστατεύσουμε λοιπόν τη στιγμή που απεδεχόμαστε αυτά τα όρια. να σα πω ειλικρινά δεν καταλαβαίνω την Επιτροπή μα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε λογικοί Ξέρουμε ότι επηρεάζει τα έντομα αυτές οι ουσίες και συγκεκριμένα του φοξαφλόρ. Θα πρέπει να αποτρέπουμε τις μέλισσες να έρχονται σε επαφή μαζί με, αυτό, ε, με το προϊόν αυτό. Ξέρουμε ότι έχει επιπτώσει την υγεία, έχει αποφασίσει ένα γαλλικό δικαστήριο να την απαγορεύσει, οπότε συνάδελφοι σας ζητώ να είμαστε λογικοί και να ακολουθήσουμε και να στηρίξουμε τους συναδέλφους, τον συνάδελφο που έχει καταθέσει αυτή την πρόταση ψηφίσματο. Πάντως οι πράσινοι θα το στηρίξουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Αν όχι, να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Μπέρεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον, ε, την συγκητρία και τα μέλη που πήραν το λόγο. Πολλά από τα στοιχεία τα οποία ήθελα να διευκρινίσω τα... μου τα πρόλαβε ο κύριος Φιέλνερ. Άρα ίσως να ακουστούν ε, κάποιες επαναλήψεις. Η πρόταση που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με το σχέδιο ε, έχει να κάνει με τα, τα μέγιστα όρια υπολοιμάτων στα τρόφιμα. Δεν έχει να κάνει με την έγκριση της ενεργούς ουσίας. Ε, σύμφωνα με τον 707 ε, του 2009. Και γι' αυτό λοιπόν η πρόθεση της εισηγήτριας να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει την έγκριση αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω ένστασης τουλάχιστον στην προκειμένη ε, πρόταση. Όπω είπε ο Σχέλνερ; η σουφοξαφλόρη δεν αποτελεί νέο νοικοϊτοειδές και δεν θα πρέπει να μπει στην ίδια κατηγορία. Η επίδραση της υποξαφλώρης στις μέλισσες εξετάζεται ήδη και θα συνεχιστεί να εξετάζεται. Το διευκρίνησε ο κ. Πότς. Και να σας απαντήσω ότι τα δεδομένα τα οποία χρειαζόντουσαν για την διαδικασία αυτή υποβλήθηκαν τον Αύγουστο του 2007 και ήδη εξετάστηκαν από τον εισηγητή και τον συνεισηγητή στην Τσεχία και η ΕΦΣΑ στην παρούσα φάση αναθεωρεί την αξιολόγηση αυτή. Και προφανώς, αν παραστεί ανάγκη να αναθεωρήσουμε την έγκριση, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε πρόταση ε, πρώιμης απόσυρσης του προϊόντος, όπω κάναμε και στην ίδια επιτροπή με άλλα νεονικοτινοειδή. Και θα ψηφίσουμε σχετικά την Παρασκευή. Άρα η αρχή παραμένει. Κάθε ουσία θα πρέπει να εξετάζεται τα σήμερα δεδομένα τα οποία έχουν συλλεχθεί για την ουσία αυτή. Δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσει τύπου όλε οι ουσίε ε, έχουν τα ίδια αποτελέσματα, ακόμα και να έχουν τα... είναι στην ίδια, στην ίδια τάξη. Γιατί όπω εξήγησα και την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμα και τα νεονικοτινοειδή ε, έχουν διαφορέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πίνακα που έχει να κάνει με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η ΕΦΣΑ, όπως είπε και ο Σχέλνερ, διευκρίνησε ότι τα προτινόμενα όρια είναι ασφαλή για την ανθρώπινη ζωή και δεν υπάρχει λοιπόν κανένας επιστημονικός λόγος να αντιταχθούμε σε αυτό. Η δικαστική απόφαση στη Γαλλία, από όσο καταλάβαμε, δεν έχει ακόμα αλευθεριστική δικαστική απόφαση, είναι σε αναστολή και είναι σε εξέλιξη η αγωγή. Η κυρία Ριβαζή διευκρίνησε ότι η Σουφουζαξαφλόρη ήταν απαγορευμένη στη ΣΥΠΑ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, έξω, όσων γνωρίζουμε. Η Αμερικανική υπηρεσία έχει εγκρίνει εκ νέου την ουσία αυτή τον Οκτώβριο του 2016. Και πάλι όμως αυτό δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη πρόταση που έχει να κάνει με τα όρια υπολοιμάτων στα τρόφιμα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταίο στοιχείο. Να σας πω ότι στο σχέδιο πρότασης αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία γραμματοδότηση στο σημείο 5 από την Επιτροπή και τις σχετικές επιτροπές και έχει λάβει ε, απορριπτικές γνωμοδοτήσεις από το Κοινοβούλιο και αυτό δεν ισχύει για την συγκεκριμένη πρόταση. Όπως σημείωσε ο κ. Φιέλνερ, ήταν σχεδόν ομώνυμη Αμα η απόφαση. Μόνο ένα κρατός μέλος αντιτάχθηκε για λόγους που δεν είχαν να κάνει με την Σουξαφλόρη. Ήταν λοιπόν ομοφωνή σχεδόν η απάντηση, ούτε στο Κοινοβούλιο απορρίφθηκε η πρόταση μας. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι και αυτό δεν στέκει απόλυτα. Συνοψίζοντας, πιστεύουμε ότι η, πρώτη η πρότασή μας συνάδει απόλυτα με τους κανόνες και τους στόχους του κανονισμού MRA, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με την ε, πιστοποίηση του προϊόντος σύμφωνα με τον 11.07.2009, 2009 αλλά προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των μελισσών και αν από τα δεδομένα που θα προκύψουν προκύψει η ανάγκη να επανεξεταστεί η σουκτοξαφλόρη, θα γίνει προφανώς κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Λέει η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα. Και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, η ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στρατηγική προσέγγιση στην ρήπανση των υδάτων με φαρμακευτικές ουσίες. Και ως συνήθως θα ξεκινήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε την κυρία Φρέτη, η οποία είναι διευθύντρια στην DG Και μετά το λόγο θα έχουν οι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο κύριε Μανφρέτη. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΕΝΒ. Είναι η πρώτη μου εμφάνιση ενώπιον της Επιτροπής σας γιατί διορίστηκα διευθύντρια τον περασμένο Φεβρουάριο 1η Φεβρουαρίου. Μόλις λοιπόν ανέλαβα τα καθήκοντά μου και είναι μεγάλη τιμή που ξεκινώ τη συνεργασία μου μαζί σας και μάλιστα για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο είναι η στρατηγική προσέγγιση για τα φαρμακευτικά. Κάτι το οποίο το ετοιμάζουμε εδώ και χρόνια ως πρόταση. Είναι νομική υποχρέωση για μας ε, και διευκρινίζεται στην οδηγία για τις ουσίες πετρεότητα. Σε κάποιε περιπτώσει η επιστημονική κοινότητα ερευνά τι επιζήμιε, ζημιογόνε επιδράσει των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον. όπω θα φαντάζετε πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μα απασχολεί πάρα πολύ και το οποίο το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και για αυτό ω Γενική Διεύθυνση περιβάλλοντό. συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με του συναδέλφου από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και με πολλές πολλές άλλες υπηρεσίε τη Επιτροπής. Τα σημαντικά μηνύματα που θα ήθελα να σα μεταβιβάσω σήμερα το πρωί είναι τα εξή. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων στην παρούσα φάση και αυτό αποτελεί κρίσιμη φάση στι ιστορικέ προετοιμασίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί σε επίπεδο υπηρεσιών έχει γίνει ήδη μεγάλο όγκο δουλειά. Έχει γίνει δημόσια διαβούλευση το 2017 μαζί με στοχευμένη διαβούλευση κάποιων ε, εμπλεκόμενων φορέων, έχουν γίνει και κάποιες μελέτες και εμείς σιγά σιγά καταρτίζουμε τα πορίσματά μας, τα ιστορικά μας πορίσματα. Σε εσωτερική, από εσωτερική άποψη προσπαθούμε να αποφασίσουμε ποιος θα είναι ο μορφότυπος των στρατηγικών αυτών εγγράφων, ποια θα είναι η χρονική στιγμή δημοσίευσης κτλ. Άρα είμαι λίγο σε μια δύσκολη θέση σήμερα το πρωί, γιατί θέλω να σας δώσω πολλές πληροφορίες και γιατί πολλά ζητήματα όμως είναι ακόμα υποσυζήτηση. Αυτό που είναι σαφές είναι το εξή. Ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να έχουμε μια ανακοίνωση η οποία θα περνούσε το μήνυμα ότι το περιβάλλον και η ανθρώπινη υγεία είναι αλληλοσυγκρούμενες ε, έννοιες και ότι θα πρέπει να διαλέξουμε το ένα ή το άλλο. Θέλουμε καταρχά να έχουμε υψηλού επίπεδου προστασία της ανθρώπινης υγείας, ενώ παράλληλα να προωθήσουμε την φαρμακευτική βιομηχανία να παράγει προϊόντα λιγότερο επιζημία για το περιβάλλον. Θα συζητήσουμε και λίγο αργότερα το θέμα της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Και στο πλαίσιο αυτό, όταν προετοιμάζαμε λοιπόν την πρόταση αυτή, αναρωτιόμασταν ήδη διάφορα για διάφορα ζητήματα, κατά πόσον θα έπρεπε να κοιτάξουμε και να συμπεριλάβουμε κάποιες παραμέτρους για τα, φαρμακο... για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του πόσιμου υδατός. Θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα. Θα δείτε ότι έχουμε συμπεριλάβει και κάποιες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα οι ενδοκρινικοί διδράκτες. Και έτσι θα ελέγξουμε τις αντικά συνέπειε και θα προσμετρούμε τον αντικτύπο όλων των στοιχείων αυτών. Εκ παραλληλού, με, στα αποστολή συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που κάνει συγκεκριμένε συστασει προ την Επιτροπή για την προετοιμασία της, οδηγία οδηγίας για το πόσιμο νερό, αποφασίσαμε να μην πάμε πολύ παραπέρα στην παρούσα φάση γιατί δεν υπάρχουν πολύ απλά επιστημονικά τεκμήρια σε ό,τι αφορά την καταναλώση φαρμακευτικών προϊόντων και κατά πόσο αποτελούν ε, κίνδυνο για την υγεία. Ε, εκ παραλλήλου, ε, μελετάμε το ζημιογόνο αντίκτυπο στο περιβάλλον και εδώ έχουμε κάποια στοιχεία και τεκμήρια για προβλήματα. Και έχουμε και τεκμήρια ότι το πρόβλημα αυτό ξεκινάει από ένα ποσοστό φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Και ήδη το 2017, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τη στρατηγική της για τον πλανήτη και την υγεία στον πλανήτη και σε ό,τι αφορά τα θέματα αντιμικροβιακής αντοχής εντόπισαμε ότι τμήμα του προβλήματος έγκυται στις ε, έλλειψη ασφάλειας σε ό,τι φορά κάποιους παραμέτρους για τα φαρμακευτικά προϊόντα σε κάποιες χώρες. Και αυτή η στρατηγική λοιπόν πρόταση θα πρέπει να καταλήξει σε κάποιες κατευθυντήριες γραμμέ για καλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρίσιμων εταίρων που παράγουν φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία στη συνέχεια διαθέτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αγορά και θεωρούμε ότι είναι η πηγή του προβλήματος. Εργαζόμαστε πάρα πολύ στενά και με τους αδέλφους από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, γιατί ένα από τα άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία εξετάζουμε είναι σε τι βαθμό θα πρέπει να αυξήσουμε τις εξάντε ε, διαδικασίε για την πιστοποίηση προϊόντων και την αξιολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων πριν την ε, πιστοποίησή τους δηλαδή. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να σας δώσω πιο πολλές λεπτομέρειες στην παρούσα φάση και φυσικά θέλω να κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό και ο Επιτροπός επιθυμεί να το προωθήσει, θέλει να το καταθέσει μαζί με τον Επιτροπό Ανδρέου Κάιτη, με τον οποίο και γίνονται συζητήσει στην παρούσα φάση και με χαρά μου θα συνεχίσω να σα τηρώ ενήμερου για οποιαδήποτε εξέλιξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει και πρόεδρο. Τώρα να συζητήσουμε το θέμα αυτό και έχω σημειώσει τα ονόματα διαφορών συναδέλφων. Η κυρία Σφαγερ Πυρίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στην Ολλανδία το θέμα αυτό είναι πολύ επίκαιρο. Και ξέρω τα θέματα επιμόλυνση του νερού από φαρμακευτικά προϊόντα στο νομοσχέδιο λοιπόν των ε, Υπουργείων το θέμα της επιμόλυνσης του νερού είναι πάρα πολύ υψηλό και επιτέλους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντηση σε γραπτή ερώτηση επιβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει σχετική στρατηγική πριν το καλοκαίρι. Το θέμα λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πιστεύει για συγκεκριμένα μέτρα σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ε, κίνητρα αλλά και υποχρεώσεις για την προστασία του νερού. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε σε επίπεδο της φαρμακοβιομηχανίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιμόλυνση καταδεικνύει σε επιφανειακά ύδατα ύπαρξη α, ανησυχητικών μικροβίων. Θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι είδους φάρμακα δημιουργούν πρόβλημα και έχουν παρουσία στα επιφανειακά ύδατα και προκαλούν πρόβλημα στα πόσιμα ύδατα, γιατί είναι Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, μας απασχολεί ιδιαίτερα στην Ολλανδία σε ό,τι αφορά την χρήση των λιμάτων και τη διάθεση των λιμάτων στην, στα νοσοκομεία στην Ολλανδία. Αυτό το άρθρο λοιπόν έχει να κάνει με την ε, α, ποιότητα των επιφανειακών υδάτων και του πόσιμου ύδατος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πέρα από τα αγροτικά μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mr. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Σέικαουτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φανταστικό νέο που επιβεβαιώθηκε ότι είναι ζωτική σημασία το όλο θέμα και για σας. Όμως ως τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φαίνεται να εργαζόταν πολύ σκληρά για να δείξει πόσο σοβαρό ήταν ε, για σας. Ε, Μα είπατε ότι είσαστε υποχρεωμένοι να το κάνετε, αλλά δεν τηρήσατε τι προθεσμίε που είχαν συμφωνηθεί. Η στατική προσέγγιση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2015 και οι νομοθετικέ προτάσει άρχισαν να βγαίνουν το 2017. Ήδη δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδειξε πόσο ε, είχε αδυναμία στο θέμα αυτό και το 2018 βρισκόμαστε να ε, προσπαθούμε να τρέξουμε πίσω από θεσμίες που συμφωνήθηκαν το 2014. Αυτά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά πραγματικά δεν καταλαβαίνω από πού προκύπτει όλη αυτή η καθυστέρηση. Τώρα μα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο σοβαρό είναι το θέμα και έρχονται τρία χρόνια αργότερα και ακόμη δεν υπάρχει στρατηγική. Ξέρω, λέτε, ότι θα είναι έτοιμη πριν το καλοκαίρι, αλλά μας έχετε γεμίσει υποσχέσεις. Δεν ε, θα περιμένουμε και κάτι πολύ καλύτερο, μα να μας εκπλήξετε. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι αυτό είναι το παρελθόν ίσως να έχει να κάνει με την καλύτερη νομοθεσία, το better regulation. Δεν ξέρω τι σημαίνει τελικά, αλλά ίσως να σημαίνει απλώς λιγότερη προστασία για τους πολίτες μας. Τώρα ας δούμε τις περιβαλλοντικές συνέπειες των φαρμακευτικών προϊόντων. Αυτό είναι το βασικό θέμα εδώ. Διότι ως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, αρνηθεί να κοιτάξει την ε, περιβαλλοντική διάσταση και τις συνέπειες των φαρμακευτικών προϊόντων τα φάρμακα είναι καλά για τον κόσμο, οπότε δεν μας νοιάζει ο περιβαλλοντικός τους αντίκτυπος. Λοιπόν, χαίρομαι που η Γενική Διεύθυνση ΕΝΒ τώρα συνεργάζεται με τους υπευθύνου για να προτείνει κάτι, αλλά ήδη κάποιες προτάσεις από την αρχή της χρονιάς πέρασαν σε ε, διοικητικές διαβουλεύσεις πού έχουν φτάσει τώρα και πού είναι η πρόταση που ασχολείται ακριβώς με, το με την περιβαλλοντική αξιολόγηση, την περιβαλλοντική μελέτη εντεκτύπου για τα φάρμακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να κοιτάξει να αυξήσει τη διαφάνεια όλε αυτέ τι αλυσίδε παραγωγή. Χρειάζεται ένα δημόσιο μητρό, όπου όλε οι τοξικολογικέ πληροφορίε και δημοσιοποιούνται και μπορεί ο καθένα να λάβει γνώση αυτών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, σα παρακαλούμε, κάντε επιτέλου τι προτάσει σα και λίγο περισσότερε λεπτομέρειε για το τι θα περιλαμβάνει η πρόταση αυτή. Γιατί και ζωτική σημασία είναι και επιτέλου είναι καιρό κάτι να κάνετε και να ε, επιτύχετε ένα αποτέλεσμα. Κάτι παραπάνω από τα λόγια που μόλι ακούσαμε ξανά. Πρόεδρο, ευχαριστούμε, κυρία Γκοντίν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έναρξη της συζήτησης αυτής για τη στρατηγική προσέγγιση και την ε, ρήπανση μόλις του νερού από τα φάρμακα είναι σημαντική. Διότι εδώ έχουμε διάφορα στοιχεία ε, που δεν ε, συμπίπτουν στις απόψεις τους και είναι από εδώ και από εκεί. Οι καταναλωτές καταγγέλουν. Οι πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει δεν είναι επαρκή. Στο 2002 η μελέτη έμπρε του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου ανείχνευσε πάνω από 80 φάρμακα στην επιφάνεια των υδάτων μιας δεκάδας ανεπτυγμένων χωρών. Αυτή τη στιγμή που η επεξεργασία, οι μονάδες επεξεργασίας των λιμάτων δεν ε, μπορούν να παλέψουν τελείως την παρουσία φαρμάκων, υπάρχουν ε, ε, προβλήματα σε, πολλές, ε, σε πολλούς συντροφορούς ορίζοντες ή σε επιφανειακά ύδατα με τη διαζεπίνη λόγου χάρη αγχολητικό που έχει ανεχνευθεί σε πολλές περιπτώσεις. Όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά στοιχεία διότι δεν μπορούμε να καταμετρήσουμε ακόμα τις άμεσες συνέπειες, τα αντιβιωτικά που χρησιμοποιούνται μαζικά στην γεωργία και την κτηνοτροφία. Ε, πλήττουν το ανασωπητικό των βιοτόπων μας. Η ορμονική αυξητικές γυναικείες ορμόνες ε, έχουν ε, ανακατευτεί με ενδοκρινικούς διαταράκτες. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφή, διότι δεν ξέρουμε τι γίνεται με τη χρόνια επίδραση, έστω και σε μικρέ δόσει αυτών των χημικών ουσιών από φάρμακα στα νερά μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζει τα επίπεδα ε, που ανησυχούν και τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ποιες, ε, ποια μέτρα θα λάβετε για να αλλάξει βάθρον το ευρωπαϊκό σύστημα επεξεργασία λιμάτων και να ασχοληθούμε με την μελλοντική διαχείριση του θέματος. Ευχαριστούμε κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και την Επιτροπή που έχει έρθει εδώ για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Απλώ να επαναλάβω κάτι σημαντικό. Η στρατηγική προσέγγιση για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα ε, είχε ανακοινωθεί ε, για τον Σεπτέμβριο του 2015 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή καθυστέρησε τουλάχιστον δυόμιση χρόνια. Θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί. Γιατί συνέβη αυτό, πείτε μας συγκεκριμένα. Γιατί να μας λέτε σήμερα, δυόμιση χρόνια αργότερα, ότι πολλά ε, σε ζητούνται εσωτερικώ. Να μα λέτε ότι δεν μπορείτε να μα δώσετε ακριβεί πληροφορίε μετά από δυόμιση χρόνια. Ε, με κάθε σεβασμό δείχνεται έλλειψη σεβασμού. Όχι μόνο προ την Επιτροπή αυτή, αλλά προ του πολίτε γενικώ και τι υποχρεώσει που αναλάβατε. Και ε, επαναφέρει το ερώτημα γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα, δυόμιση χρόνια αργότερα. Το λέω διότι είναι γνωστό ότι τα κατάλοιπα από φάρμακα και έχουν ανοιχνευτεί στα επιφανειακά ύδατα και σε υδροφόρους ορίζοντες και σε υπόγεια ύδατα, σε πόσιμο νερό ε, παντού σε πολλές χώρες παγκοσμίω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εμπειρογνώμονες και ακόμη και οι εμπειρογνώμονες στο ΙΕ λένε ότι έχουμε ένα, ένα παγκόσμιο πρόβλημα μόλις από φάρμακα και πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσον μπορεί να πετούνται τα φάρμακα στο περιβάλλον και το τι θα κάνουμε με τον κύκλο ζωή των φαρμάκων, την ε, αποκομιδή του και την αποθήκευση. Πρέπει λοιπόν σήμερα να σκεφτούμε ακριβώ τι θέλουμε να κάνουμε δυόμιση χρόνια μετά την αναγγελία για τη στρατηγική προσέγγιση. Και αυτό πρέπει να συνδυαστεί με το σχέδιο δράση για την παρακολούθηση τη αντιβιωτικ... αντίδραση στα αντιβιωτικά τη ανθεκτικότητα στα βακτήρια λόγω τη διάδοση των αντιβιωτικών, κάτι που έχει μακροχρόνιε επιπτώσει στην υγεία. Είναι απαράδεκτο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ακολουθεί τη διαδικασία που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και ναι, περιμένουμε ο δικό χάρτη να δημοσιευτεί αμέσω, για να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα τη ρήπανση από φάρμακα αμέσω. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα πει πότε, πότε θα έχουμε αυτή τη στρατηγική προσέγγιση. Τι σα εμποδίζει να την ε, σχεδιάσετε και ποια είναι αυτά που εσωτερικώς ακόμα συζητάτε σε επιρρησιακό επίπεδο. Περιμένουμε και την πρόταση και τη στρατηγική προσέγγιση διακαώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φόλκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Τάλη. Όντως. Εδώ και καιρό περιμένουμε τα στοιχεία αυτά. και είχα και μια σχετική εκδήλωση στο Κοινοβούλιο και να σας πω ότι οι 15 ενδιαφερόμενοι όταν ε, έμαθαν για τις πρώτες ε, ενδείξεις για το τι θα συμπεριβαλλοντούσαν, τι θα συμπεριβαλλοντούσαν, ε, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά. Και άρα υπάρχει μεγάλη αγωνία. Και επιτέλους χρειαζόμαστε κάτι συγκεκριμένο για να δουλέψουμε. Γιατί αυτό το πρόβλημα και το είπαν οι προηγούμενοι ομιλητέ, είναι ένα θέμα το οποίο ταλωνίζει τους πολίτες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όντως, πιστεύω ότι είναι ένα τμήμα του πακέτου θα πρέπει να εστιαστεί σε θέματα διευκρίνησης, διελεύκανσης, γιατί είναι σημαντικό να κοιτάξουμε και στα ήδη χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά προϊόντα πώς επηρεάζουν τα έδατα. Δηλαδή υπάρχουν φάρμακα τα οποία μπορούν να φιλτραριστούν πολύ καλά στο πόσιμο νερό, αλλά υπάρχουν και άλλα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για ακριβώς τον ίδιο σκοπό και δεν φιλτράρονται στο νερό. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να προσέξουμε να χρησιμοποιούνται προϊόντα τα οποία φιλτράρονται καλύτερα. Αυτό λοιπόν πιστεύω θα αποτελεί τμήμα του πακέτου για τη μείωση ε, των υπολοιμμάτων τέτοιων ουσιών ε, στο περιβάλλον ε, είναι, θα πρέπει να είναι πολύ καλύτερη. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μια ερώτηση η οποία σχετίζεται και με την αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Όλοι ξέρουμε ότι οι εταιρείε υδροδότησης θα αναγκαστούν σύντομα να εισαγάγουν ένα τέταρτο επίπεδο καθαρισμού του νερού. Και θα είναι κοστοβόρο και δεν θέλω αυτό το κόστος να μετακυλιστεί στον καταναλωτή. Πώς λοιπόν θα εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εφαρμογή της αρχής του ΡΥΠΕ πληρώνει σε αυτά τα σημαντικά θέματα. Επίσης, κατά πόσο υπάρχει διαδικασία, παρακαλώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πείτε μου, για την παρακολούθηση ε, πολυεντακτικών ε, μικροβίων στο νερό. Γιατί θα πρέπει να έχουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει. Ευχαριστώ ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συναδελφοί, βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρυθμό εργασίας της Επιτροπής όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα φαρμακευτικά. Και το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και καιρό. Και ξέρουμε ότι μετά το μεγάλο boom στην ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα αυτό είναι πιο έντονο. Ξέρουμε ότι το θέμα των αντιβιωτικών ήταν κάτι το οποίο δεν αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν επειδή τα χρησιμοποιούμε τα αντιβιωτικά πολύ περισσότερο σήμερα. Ξέρουμε ότι αυτές οι ουσίες ξέρουμε ότι διαταράσσουν την ορμονική ισορροπία τα αντιβιωτικά και αυτό όντως αποτελεί πρόβλημα. Οπότε θα ανέμενα από την Κομισιόν καταρχάς να προσπαθήσει να εντοπίσει τις πηγές από τις οποίες προέρχονται όλες αυτές οι ουσίες. Δηλαδή, να δούμε τελικά πώς καταλήγουν αυτά τα φάρμακα στα ύδατα και ποιος είναι υπεύθυνο γι' αυτό. Ευθύνονται οι παραγωγοί Ίσως για λόγους παραγωγής στα εργοστάσια να υπάρχει ένα κλειστό κύκλωμα και με αυτόν τον τρόπο να απέτρεπε τέλο πάντων την διάχυσή του ε, στα ύδατα, ώστε να μην φτάνουν και στα πόσιμα ύδατα και πρέπει εδώ να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχει κάποια, κάποια τέτοια λύση. Τώρα, όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας και τα οποία θέλουμε να πετάξουμε, έστω και αν ε, δεν τα έχουμε τελειώσει, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτά βλάπτουν το περιβάλλον, βλάπτουν επίσης και τα ζώα όταν διατίθεται στην ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι επίσης ε, σοβαρό πρόβλημα. Οπότε, Πρόεδρε, στον τριμερή διάλογο για τα φαρμακευτικά έχουμε έλθει σε αδιέξοδο για αυτά τα ζητήματα. Και νομίζω ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν θέλουμε και δεν ξέρουμε ακριβώς μάλλον τι θέλουμε να κάνουμε με αυτά τα φαρμακευτικά απορρίμματα και τις επιπτώσεις που έχουν στην υγεία μας και στο περιβάλλον. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα, αλλά υπάρχει ένας οδικός χάρτης. Αν αυτός ο οδικός χάρτης δεν επαρκεί, το θα πρέπει να φτιάξουμε έναν άλλο το ταχύτερο δυνατό. Και βλέπω ότι δυστυχώς η Κομισιόν δεν έκανε αυτό που περιμέναμε. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει τεράστιες επιπτώσεις. Βεβαίως χαιρετίζουμε την αφύπνιση, να την πω έτσι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ίσως να κοιμόταν μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα σε πέντε χρόνια να μην ξαμιλάμε αυτά τα ζητήματα. Οπότε το ερώτημα παραμένει. Έχετε εντοπίσει τις πηγές αυτών των προβλημάτων. Ποιε είναι οι πηγές μόλυνσης των φαρμακευτικών προϊόντων στο περιβάλλον και στα ύδατα και ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να να εξετάσουμε δηλαδή πόσο οφείλεται στην γεωργική παραγωγή, πόσο οφείλεται στη μόλυνση από φάρμακα που προέρχονται από τα σπίτια. Θα πρέπει να δούμε επίση πόσο κοστίζει η προσπάθεια αυτή ώστε να εξαλείψουμε τέλο πάντων τα κατάλοιπα αυτά από τα φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον και στην υγεία μα. Γιατί θα έχει κάποιο κόστο και φαντάζομαι το κόστο θα είναι σχετικά υψηλό. Οπότε καλύτερα να επαγρυπνούμε όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέω ο Σταντάν. Ευαίσθητο και επίμαχο αυτό το θέμα. 50% των αποβλήτων των φαρμακευτικών προϊόντων έδειξε μια μελέτη στη Γαλλία ότι προέρχονται από τα νοσοκομεία. Η Κομισιόν διαθέτει αντίστοιχα, αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Εμείς όλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και κάποια χρόνια Έχουμε προωθήσει τους ε, σταθμούς βιολογικού καθαρισμού. Αυτή τη στρατηγική για τους σταθμούς βιολογικού καθαρισμού θα την αναθεωρήσετε και για την ανθρώπινη υγεία θα ξανασυζητήσουμε την οδηγία για το πόσιμο νερό εν ώψη των στοιχείων που διαθέτει η Κομισιόν. Μήπως θα έπρεπε λοιπόν να πάμε παραπέρα στα πλαίσια της οδηγίας για, τα, για το πόσιμο νερό και αν ναι, με ποιες παραμέτρους. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι όπως είπαμε προηγουμένως οι σταθμοί βιολογικού καθαρισμού δεν φιλτράρουν κάποια στοιχεία, κάποια συστατικά των φαρμάκων. Οπότε μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και στην έρευνα πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε μια έρευνα σωστή ώστε να καταλήξουμε σε μια σωστή μέθοδο ώστε να σταματήσουμε ακριβώς την διάχυση αυτών των προϊόντων στο πόσιμο νερό. Ευχαριστώ. Μετά την επεξεργασία στους σταθμούς καθαρισμού, θέλω να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρο. Ε, κάποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Αλλιώ η κυρία Μανφρέντι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Μανφρέντι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω φαντάζεστε, ε, δεν έχω πρόθεση να δείξω ασέβεια στην πρώτη μου παρθενική μου εμφάνιση στην Επιτροπή σας. Είμαι ευσεβής και δεν φυσικάζω. Κάθε άλλο. Ήθελα να δείξω ακριβώς σεβασμό για το γεγονό ότι υπάρχει ακόμα μια ενεξελίξη εσωτερική διαδικασία. Εμείς πάντως κάναμε ό,τι έπρεπε και να σας αναφέρω κάπως περισσότερο το τι προτιθέμεθα να κάνουμε. Η στρατηγική λοιπόν θα βασίζεται σε έξι βασικούς πυλώνες που αφορούν διάφορα συστατικά στοιχεία. Γιατί εμείς θέλουμε εδώ να εξετάσουμε το σύνολο του κύκλου ζωής της παραγωγής των φαρμακευτικών προϊόντων. Παραγωγή, έγκριση, διάθεση, απόρριψη. Οπότε θα πρέπει να είμαστε σε θέση, και αυτή την πρόθεση έχουμε, να, να παρεμβαίνουμε στην κάθε φάση χωριστά, ώστε να έχουμε στην αγορά λιγότερο βλαβερά φαρμακευτικά προϊόντα. Αυτό όμως απαιτεί και μια αλλαγή νοοτροπίας. Αλλαγή νοοτροπίας σε επίπεδο χρηστών και γιατρών που τα συνταγογραφούν σε συνεργασία βέβαια και με την φαρμακοβιομηχανία που τα παράγει. Κάποιοι ζητήσατε περισσότερο ακριβείς ε, πληροφορίες σε σχέση με τις πηγές αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων. Υπάρχει μια συνεχής εποπτεία και γνωρίζουμε και πρέπει να ξέρετε κι εσείς ότι ανανεώσαμε πρόσφατα το κατάλογο υπό επιτήρηση που συμφώνησαν να συγκροτήσουν χώρε μέλη και να τοποθετήσουν τι ουσίε οι οποίε θα πρέπει να, να ελεγχθούν και να αποπτευθούν για κάποιο χρονικό διάστημα και υπάρχουν ουσίε όπω το αμοξίλιουμ και το τσιπροφλοξασίν. Αυτέ είναι υπάρχουσε ουσίε οι οποίε ήδη βρίσκονται σε αυτόν τον κατάλογο προ επιτήρηση. Αυτή λοιπόν δουλειά που συνεχίζεται με τους ε, συναδέλφους των ε, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, τις αρχές των υδάτων, τα Υπουργεία Υγείας κλπ. Και αυτό βέβαια με οδηγεί στην απάντηση στο κέριο ερώτημά σας. Γιατί, γιατί, γιατί, γιατί άργησε η Κομισιόν, γιατί δεν τηρήσαμε την προθεσμία στο μέτρο του δυνατού, όπως λέει η οδηγία, έτσι, του 2015. Η απάντηση είναι επειδή ακόμα συλλέγουμε πληροφορίες και θέλουμε να υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να έχουμε μια σωστή στρατηγική. Θέλω όμως να σας ενημερώσω ότι θα είναι μια ολιστική, συνολική στρατηγική η οποία θα προτείνει περαιτέρω βήματα έρευνας και διερεύνησης. Να μιλήσω για τους έξι πυλώνες που ανέφερα. Ο πρώτος πυλώνας θα εξετάζει ακριβώς το κατά πόσο μπορούμε να αυξήσουμε την επίγνωση για τη μη ουσιώδη χρήση για τα ανθρώπινα και κτηνοτροφικά φάρμακα ώστε να καθησυχαστούμε πραγματικά ότι όντως εξετάζουμε το τι γίνεται και με τη χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων για τη θεραπεία των ζώων σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και παρακολουθώντας βέβαια στενά τις, τις διαπραγματεύσεις που γίνονται στα πλαίσια του κοινοτροφικού πακέτου. Ο δεύτερος πυλώνας αποβλέπει στην υποβολή συγκεκριμένων μέτρων για να τονώσουμε την ανάπτυξη και την χρήση από τους καταναλωτές πιο πράσινων φαρμακευτικών προϊόντων και αντίστοιχη παραγωγής τους. Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με το δεύτερο, η ενίσχυση δηλαδή της χρήσης ε, διαδικασιών αποτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου πριν τεθούν τα φαρμακευτικά προϊόντα στην αγορά. Τέταρτος πυλώνας εξετάζουμε τα μέτρα τα οποία αποβλέπουν στην χρήση της απόρριψης αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων και βελτίωση της διαχείρισής τους. Πέμπτος πυλώνας θα διευρύνει και θα επεκτείνει τις δράσεις μας σε συνεργασία στενή με τις αρχές, τους εμπλεκόμενους, τα κράτη ώστε να ενισχύσουμε ακριβώς την εποπτεία σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στη στρατηγική θέλουμε να εντοπίσουμε κάποια hot spots και μέρη όπως νοσοκομεία όπου εκεί θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, τέλος, υπάρχει ένα κεφάλαιο που αφορά τις ελλείψεις στις γνώσεις μας, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν με περαιτέρω έρευνα. Φαντάζεστε σε όλα αυτά ότι η δουλειά που γίνεται στον τομέα των υδάτων, όπου έχουμε κάνει μια εκτενή αξιολόγηση της οδηγίας για τα αστικά ύδατα και την επεξεργασία τους, αυτό είναι σημαντικό και πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε μια δημόσια διαβούλευση, όπου θα δούμε ότι οι συγκεκριμένα ερωτήματα ακριβώς αφορούν το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές παραμέτρους για να διασφαλίσουμε καλύτερη επεξεργασία των εδάτων και σε σχέση με τα φαρμακευτικά προϊόντα αλλά και τα μικροπλαστικά, τα οποία είναι βεβαίω και αυτά μια νέα πρόκληση. Αυτή η δουλειά λοιπόν κουμπώνει πολύ ωραία με την ε, δουλειά που γίνεται με τις οδηγίες που αφορούν τα ύδατα και προσπαθούμε επίσης να δούμε κατά πόσο μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα έγγραφο από την Κομισιόν με όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί όταν θα ξεκινήσουμε όλα αυτές τις ε, δράσεις, θα δούμε πώς όλα αυτά θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τη δουλειά που θα κάνει η Κομισιόν για τον έλεγχο της συνολικής ισχύς και αποτελεσματικότητα όλων αυτών των κανόνων που υπάρχουν και των νομοθεσιών. Δεν ξέρω κατά πόσο απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Αλλιώς, Πρόεδρε, παρακαλώ, πείτε μου. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Καλά, το δημόσιο μητρό. Δεν το σχολιάσατε για τις πληροφορίες από τις περιβαλλοντικές τοξικολογικές μελέτες. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Έκατ που το επαναφέρετε το σημείο αυτό. Κυρία Μανφρέντε, αν έχετε τώρα μια απάντηση. Ναι. Οι συνάδελφοι που είναι ειδικοί επί του θέματος και το μελετούν λένε ότι αυτό είναι μέρος του κεφαλαίου που θα κοιτάξουμε να υπάρξει αύξηση της διαφάνειας προς την ενημέρωση των καταναλωτών. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να περάσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Μόλις η στρατηγική υιοθετηθεί να απαντήσουμε στη συγκεκριμένη ερώτηση με περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βεβαίως, το Δημόσιο Μητρό είναι μέρος ε, της όλης προσπάθειας διαφάνειας ή τέλο πάντων επίτασης της διαφάνειας. Ε, έτσι, ε, ολοκληρωνεται τη συζήτησή μας και περνάμε στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την κυρία Μανφρέντι και πάλι, για την υλοποίηση της διαδικασίας για το περιβάλλον και την υγεία. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις εδώ. Και να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις για την υπάρχουσα νομοθεσία. Θα οργανωθούμε σε ομάδες θεμάτων, σε κλάστερ θεμάτων και η κυρία Μανφρέντι θα μπορεί να απαντήσει στους θέτουν ερωτήσεις για να ακολουθήσουν οι επόμενοι. Πρώτο θέμα, συμμόρφωση και ένδικα μέσα για τη χρήση. Κυρία Μανφρέντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό έχει να κάνει με την πρότασή μας για τον αναδιατύπωση της οδηγίας για τα ύδατα, στο άρθρο 12 της πρότασης υπάρχει μια πρόταση που λέει ότι τα κράτη-μέλη αυτομάτως θα εξετάζουν την αδυναμία να σεβαστούν τα κατώτατα όρια που ε, αναφέρονται και στο παράρτημα ως ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Η πρόταση αυτή σημαίνει ότι η προσφυγή ή τέλο πάντων μάλλον η προσπάθεια αποκατάσταση που ελπίζουμε να αναλάβουν τα κράτη-μέλη σε τέτοιε περιπτώσει. δεν θα καταλήξουν σε απαγόρευση κατάποσης του ύδατος. Ίσως πρέπει να δοθούν ε, συμβουλές σε συγκεκριμένε ομάδες του πληθυσμού, να μελετηθούν τα αίτια, να εκδοθούν κάποιες ειδοποιήσεις, να αναλυθούν μέτρα που δεν είναι πρώτα το τελευταίο έσχατο μέτρο που μπορεί να αναλυφθεί. Αυτό είναι παράπλευρη συνέπεια των όσων αναφέρει το άρθρο 4 της οδηγίας, όπου ξεκάθαρα αναφέρεται ότι υπάρχει γενικευμένη υποχρέωση για τα κατημέλη... να σεβαστούν τις τιμές των ε, παραμέτρων στο παράρτημα, καθώς σκοπός της συνολικής πρότασης είναι να υπάρξει ε, καλή ποιότητα για την ανθρώπινη υγεία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε εδώ πιστοί στον αρχικό στόχο της οδηγίας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πόσιμου ύδατος ε, σε μη πλήρη συμμόρφωση με όλα τα σημεία της πρότασης, άρα αδυναμία συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσει. μπορεί να οδηγήσει ενδεχομένως σε κινδύνους υγείας. Ξέρετε ότι τις παραμέτρους της ετοιμάσαμε σε στενή συνεργασία με τα Διεθνή Οργανισμό για το Νερό. Θεωρούμε λοιπόν ότι το κείμενο είναι πολύ σωστά εξισορροπημένο προ αυτό το σημείο, αλλά ευχαρίστω να συνεργαστούμε περαιτέρω μαζί σα. Πρόεδρο, απαντήσατε στην ερώτηση του κυρίου Μάντλ. Θέλει ο κύριο Μάντλ να ζητήσει διευκρινήσει, κάποιο άλλο συνάδελφο. Όχι, όχι. Ωραία. Επόμενο θέμα. Παρακολούθηση της ποιότητα των δάτων. Από τον κύριο Μάντλ, τον κύριο Φλόρεν, τον κύριο Πότς το ερώτημα, την κυρία Μίλλερ και τον κύριο Μπόλαν. Πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το θίξαμε λίγο και στην προηγούμενη συζήτηση. Είναι γεγονός ότι βάσει της ισχύουσας οδηγίας του 98 δεν έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις για τα φάρμακα, άρα δεν υπάρχουν και δεδομένα από την παρακολούθηση του τι γίνεται για τα φάρμακα στην οδηγία αυτή, βάσει της οδηγίας αυτής. Όμως το θέμα των φαρμάκων στο πόσιμο νερό έχει αναλυθεί σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να δούμε κατά πόσον θα αναθεωρηθούν και σχετικές ε, τιμές που αναφέρονται στην οδηγία. Η τελική σύσταση του ΠΟΗ λέει ότι θα ήταν ε, ανάρμοστο να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα φάρμακα στο παροτιμένα της οδηγίας αυτή τη στιγμή, ε, ενώ αναγνωρίζει ότι κάποια συνολική και γενική παρακολούθηση πρέπει να υπάρξει. Το εργαλείο μέσα του οποίου η πρότασή μας λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένε τιμέ για τα φάρμακα είναι μέσω του άρθρου 8, αυτό που ονομάζουμε ε, αξιολόγηση κινδύνου. Διότι, όπω τα γνωρίζετε, στο πλαίσιο του άρθρου αυτού, τα κράτη-μέλη πρέπει να εκπονήσουν συγκεκριμένη μελέτη ανάλογα με το σημείο ε, καθαρισμού, επεξεργασίας από το οποίο παίρνουν το νερό για να κάνουν τη μέτρηση. Πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη και αυτό το γεγονός. Α σκεφτούμε λοιπόν την περίπτωση που ένα ποτάμι περνάει κοντά από ένα νοσοκομείο. Είναι ένα hot spot είναι επίσης ε, ανάλογο το αν υπάρχει κοντά ένα χημικό εργοστάσιο που φτιάχνει φάρμακα. Εκεί το νερό που περνάει θα περιέχει ενδεχομένω περισσότερες επικίνδυνες χημικές ουσίες. Η ανάλυση του νερού από αυτό το συγκεκριμένο σημείο θα ε, οδηγήσει στην ε, αναγκαστική λήψη περισσότερων μέτρων. Εδώ η αναθεωρημένη πρόταση προβλέπει τρεις παραμέτρους που έχουν εντοπιστεί και πάλι σε συνεργασία με τους συναδέλφους του ΠΟΗ. Έχουν θεωρηθεί σημαντικές παράμετροι για την ενδεχόμενη παρουσία ενδοκρινικών διαταρακτών, κάτι που έχει άμεση σχέση με την παρουσία φαρμάκων στο νερό. Η μπισφονελ, ένα του μπισπροφενήλ και άλλη μία ουσία νονιλφενόλ πρέπει να βελτιώσω τις επιστημονικές μου γνώσεις ε, ως προς το θέμα. Εδώ είναι πολύ χαμηλές οι αξίες για τις παραμέτρους αυτές. Και εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται με την παρουσία των ουσιών αυτών στο πόσιμο νερό. Όπως με το συνολικό μηχανισμό της οδηγίας, ο πάροχος, ε, ο υδροδοτικός, πάροχος υδροδότησης θα πρέπει να κοιτάξει πώς θα αντιμετωπίσει την παρουσία των ε, τιμών αυτών και θα γίνει εξέλιξη κινδύνου ώστε στη συγκεκριμένη περιοχή μετά από έλεγχο να μην υπάρχουν πλέον αυτές οι αξίες. Ελπίζω ότι απήντησα στις βασικές ανησυχίες των χαξιότιμων βουλευτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα να ρωτήσω αν θέλετε να κάνετε άλλες ερωτήσεις, κατά πόσο σας ικανοποίησε η απάντηση που λάβατε. Κύριος Ποπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τους ενδοκρινικούς διδαράκτες, δύο ερωτήσεις έχω να κάνω. Θα συμφωνούσατε ότι μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά το κόστος σημαίνει μέτρα για την προστασία των υδάτων βάσει της προστασίας ε, ε, των υδάτων και της αρχής ε, του Ρηπένα και χωρίς, ε, ότι χωρίς σαφή κατανομή ευθυνών αυτή η νέα πρόταση θα καταλήξει να έχει απλά πιο υψηλό κόστος για τον καταναλωτή χωρίς να έχει απαραίτητα σε αποτέλεσμα καλύτερη ποιότητα. Τρίτη ερώτηση για τα μικροπλαστικά. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι γίνεται και τι θα γίνει στο μέλλον, ε, αν υπάρχουν μερικές πρωτοβουλίες για αξιόπιστες ε, μεθόδους ε, ελέγχου σε ό,τι αφορά την ύπαρξη μικροπλαστικών στα ύδατα. Και τι προγραμματίζει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι θα υπάρξουν οριστικές εκθέσεις για τα χημικά κοκτέιλ και την επίδραση στην ανθρώπινη υγεία και σε ό,τι αφορά τις ορευτικές ουσίες. Ευχαριστώ και το ξύνα. Η κυρία Μίλλερ. Και εγώ δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη με τις απαντήσεις. Είμαι σκιώτης εισηγήτρια από την Άλντα. Και ήμουν σε θέση δημοτικών συμβουλίων όπου είχαμε την αίσθηση τη ευθύνη που έχουμε στον πολίτη απέναντι σε ό,τι αφορά τα πόσιμα είδοντα. Αυτές οι παράμετροι λοιπόν, εισαγωγή ενδοκρινικών διαταρακτών προκαλεί μεγάλα προβλήματα. Γιατί πιστεύω, όπως και οι προηγούμενοι ότι το κόστος τελικά θα μετακυλιστεί στον τελικό χρήστη και θα είναι υπέραγκο οι δοκιμασίε για το νερό. Τελικά, και τα αποτελέσματα. Πώ εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι έχουμε εκτάσεις προστατευμένων υδάτων, όπου θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα όρια. Και στη συνέχεια να τη χάνουν εμπορίας. Και εδώ λοιπόν έχουμε δυνατότητα να διαθέσουμε, να δώσουμε ελευθερία στα κράτη-μέλη. Επίσης, αυτή η προσέγγιση βάσει κινδύνου του 2015, πώς τελικά εφαρμόστηκε στα κράτη-μέλη, έχετε να μας δώσετε κάποιο feedback. Καταλαβαίνω το πρόβλημα της ε, χρήσης αναγκαστικά φίλτρων, άνθρακα για την ε, ποιότητα του νερού κτλ. Αλλά αυτό συνεπάγεται και τελείω μεγάλο κόστος. Ε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή το refit στο άρθρο 10, διαπιστώσαμε ότι δεν πετύχαμε το στόχο μας. Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται σε λυπή εφαρμογή στα κράτη-μέλη ή έχει να κάνει με το ίδιο το άρθρο είναι προβληματικό από μόνο του. Άλλος κανείς, λέει πρόεδρος. Ο κύριος Ζόφουλη. Ehm, <clears throat> ναι, και εγώ ήθελα να γυρίσουμε σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, χημικές ουσίες που δεν είναι παρούσες στη φύση που βρίσκουμε σε κάποια αποθετικά προϊόντα στην περιοχή του Βένετο στην Ιταλία είχαμε μια μεγάλη μόλυνση από αυτές τις ουσίες με ποσοστά στο αίμα του πληθυσμού 350.000 άτομα σε διάφορες επαρχίες όπως τη Βερόνα, Πάντοβα, Βιτσέντσα κτλ. Πολύ υψηλή λοιπόν παρουσία των νησιών αυτών στο ανθρώπινο σώμα και παραμένουν εκεί 4 με 8 χρόνια μέχρι να εξαλειφθούν. Για πρώτη φορά λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο 1β του παραρτήματος καθορίζονται όρια για αυτές τις ουσίες και θα ήθελα να μάθω ακριβώς με ποια κριτήρια τέθηκαν αυτά τα όρια γιατί θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ακόμα αυστηρότερα όρια και μάλιστα οι τοπικές αρχές στο Βενέτο μετά από αυτή την υπόθεση καθόρισε όρια σχεδόν μηδενικά. Εμείς αντίθετα προβλέπουμε όρια πιο έψηλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρώτα ευχαριστώ. Στην πρόταση του κειμένου έχει αφαιρεθεί το άρθρο που αφορά τις παρεκκλήσεις φαίνεται οι χώρες να είναι προσιλωμένες στην διατήρηση αυτής της πιθανότητας μιας παρέκκλησης για διάφορους λόγους, Έχουμε και τυχαίους. Η Κομισιόν μας είπε ότι πρόσφατα είχαμε διάφορες παρεκκλήσεις και ποιοι ήταν οι στόχοι αυτών των παρεκκλήσεων και ποιος ήταν ο λόγος των παρεκκλήσεων αυτών. Και μετά προτείνεται κάποιες νέες παραμέτρους. Θα χρειαστεί χρόνος ώστε όσοι διαχειρίζονται αυτά τα δίκτυα να προσαρμοστούν Μήπως λοιπόν θεωρείται απαραίτητο ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιο χρόνο πριν ε, αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα αυτές οι απαιτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κυρία Μανφρέντι, έχετε κάποιες άμεσες ερωτήσεις για αυτό το θέμα, αλλά επίσης έχετε και την τοποθέτηση του κύριου Νταντέ για τις παρεκκλήσεις. Αφού ολοκληρώσουμε το τωρινό θέμα, μετά να πάμε και στις παρεκκλήσεις, αν συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Ευχαρίστω, ευχαρίστω. Ναι, να προσπαθήσω πρώτα να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Μίλλερ για το άρθρο 10 τη τρέχουσα οδηγία που φαίνεται ότι δεν έχει πετύχει το στόχο του. Να διευκρινίσω ότι η αναθεώρηση τη οδηγία για το πόσιμο νερό πραγματικά περιλαμβάνει αυτό το νερό, το, αυτό το άρθρο και το θεωρεί αποτελεσματικό. Γιατί αφήνει περιθώριο στις, χώρε μέλη να καθορίσουν τα απαραίτητα μέτρα τα οποία δεσφαλίζουν ότι τα υλικά τα οποία έρχονται σε επαφή με τα ύδατα τηρούν τα επίπεδα ασφαλείας για την ανθρώπινη υγεία. Και όπως ξέρετε, αυτό οφείλεται στο ότι σήμερα η βιομηχανία που παράγει αυτά τα υλικά αντιμετωπίζει σημαντικό διοικητικό φόρτο, επειδή ακριβώς θα πρέπει να αναζητήσουν διάφορες άδειες και εγκρίσεις για να έχουν αδειοδότηση σε όλη την Ένωση, με κόστος 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό οδηγεί επίσης βεβαίως και στο, στη δομή και την διατύπωση αυτού του άρθρου που αφορά την εφαρμογή στις χώρες μέλη. Επειδή κάποιες χώρες μέλη απαιτούν επιπλέον δοκιμές πριν τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά. Για αυτούς τους λόγους και βεβαίως σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους που έχουν να κάνουν με αυτά τα προϊόντα. Προτείνω λοιπόν την αναδιατύπωση για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτό το γεγονός και να διευκρινίσουμε ότι μέσω αυτού του κανονισμού θα πρέπει να αναπτύξουμε προδιαγραφές για τις δοκιμές αυτών των σημαντικών υλικών που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Θα θέλαμε βεβαίως εδώ να διευκολύνουμε την αδειοδότηση σε όλη την ενιαία αγορά, αποφεύγοντας βέβαια την επικάλυψη δοκιμών, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις, στα, στις υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Ήδη χρησιμοποιούμε κάποια προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και που προχωρούν γρήγορα και θέλουμε το φάκελο αυτό να τον ολοκληρώσουμε σύντομα μαζί με τους συναδέλφους ώστε να πετύχουμε ακριβώς υψηλή υγειονομική επίδοση αυτών των υλικών. Έχουμε και συζητήσεις στο Συμβούλιο που αφορούν τα ζητήματα αυτά. Και να επωφεληθώ τη ευκαιρία για να σας ενημερώσω ότι οι συζητήσεις στο Συμβούλιο προχωρούν καλά. Έχουμε δέσμευση από τη Βουλγαρική Προεδρία να προχωρήσουμε με το φάκελο αυτό και βασιζόμαστε βέβαια και στην δική σας συνεργασία γι' αυτό. Για τον κύριο Τσόφολη για αυτό που έθιξε να πω για αυτές τις ουσίες που ανέφερε και τον κίνδυνο που αποτελούν για την ανθρώπινη υγεία. Ξέρετε ότι η Κομισιόν αποφάσισε να περιλάβει αυτές τις ουσίες ως μια νέα παράμετρος εποπτείας για το πόσιμο νερό. Δεν υπήρχε μέχρι τώρα στην υπάρχουσα οδηγία. Θεωρούμε ότι πραγματικά εδώ θα πρέπει να ακολουθήσουμε με φιλόδοξη προσέγγιση, γιατί θα πρέπει να θέσουμε ένα νότατο όριο για όλη την ομάδα αυτών των ουσιών και για κάθε μεμονωμένη ουσία χωριστά. Και αυτό επειδή θέλουμε να αποφύγουμε το ότι κάποιες ουσίες θα αντικαθίστανται από κάποιες παρόμοιες με παρόμοια βλαβερά αποτελέσματα όπως συνέβη, όπως γνωρίζετε στις κάτω χώρες πρόσφατα όπου συγκεκριμένες ουσίες αυτού του είδους, το PFOA, αντικαταστάθηκαν από τις ουσίες Gen X, οι οποίες βεβαίως προκαλούν παρόμοιες βλάβες. Βάσει λοιπόν της αρχή της προλήψεως θα ρυθμίσουμε όλες αυτές τις ομάδες ουσιών με αξίες 0,1 χιλιοστογραμμάρια αναλύτρο για κάθε μία από αυτές τις ουσίες και 0,5 για όλες τις ουσίες στο σύνολο των, της ομάδας αυτών των ουσιών. Βεβαίω αυτέ ίσω να είναι κάπω υψηλότερε ω αξίε από αυτέ που ισχύουν στην Βρετανία ή στην Σουηδία. Οπότε ω Ευρώπη θα έπρεπε να έχουμε μια νέα προσέγγιση. Επίση αυτά που είπε ο κύριο Νταντάν για τι παρεκκλήσει. Γιατί εμεί ε, διαγράψαμε το άρθρο 9 από την τωρινή οδηγία για το πόσιμο νερό και ποια είναι η θέση μας σε σχέση με τη λειτουργία αυτού του άρθρου και τις πολλές παρακλήσεις τις οποίες είδαμε να υπάρχουν. Γνωρίζετε ότι υπό το άρθρο αυτό οι χώρες μέλη οφείλουν να υποβάλουν εκθέσει από τη δεύτερη παρεκκλήση και μετά. Υπάρχει μια περίοδος ε, τριετίας όπου δεν είναι υποχρεωμένε να υποβάλουν εκθέσει, Έχουμε ένα ε, συνολικό αριθμό παρεκκλήσεων που έχουν εφαρμοστεί λόγω της οδηγίας σε όλη την Ευρώπη. Παρόλα αυτά, έχουμε και κάποια γενική εικόνα και να σας πω ας πούμε ότι το 17 η Κομισιόν έλαβε ένα αίτημα για μια τρίτη παρέκκληση με μια παράταση 9 ετών την οποία απέρριψε το αίτημα απέρριψε. Και είχαμε και μέχρι τώρα 10 αιτήσει για πρώτες και δεύτερες παρεκκλήσεις. Θεωρούμε ότι στη φάση αυτή, τόσα χρόνια μετά από την θέση σε ισχύ της οδηγίας για το πόσιμο νερό, οι παρεκκλήσεις δεν αποτελούν πια ένα κατάλληλο εργαλείο. Ήταν ίσως κατάλληλες στην αρχή της εφαρμογή της οδηγίας, επειδή ήταν απαραίτητο να δώσουμε στις χώρες μέλη επιπλέον χρόνο για να πετύχουν τις ε, αξίες, τη παραμέτρους που είχαν καθοριστεί. Όμως τώρα που έχουμε την 15 αιτία, θεωρούμε ότι είναι παροχημένες οι παρεκκλήσεις και αδικαιολόγητες μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε και δεκτικοί σε σχέση με τα επιχειρήματα του κυρίου Ευρωβουλευτή και να ευχαριστήσω βεβαίω και τον συντάκτη για την θαμάσια συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Είμαστε λοιπόν δεκτικοί για το ενδεχόμενο ύπαρξης μεταβατικής περιόδους περίοδου ώστε να βοηθήσουμε τις χώρες οι οποίες χρειάζονται κατάλληλο χρονικό διάστημα για να πετύχουν τις αξίες. Αυτό συζητείται σε επίπεδο συνομοθετών και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους επιτρέψουμε να πετύχουν έναν καλό συμβασμό σύμφωνα με τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Δηλαδή, υψηλή προστασία της ανθρώπινης υγείας και εμπιστοσύνη των καταναλωτών όσον αφορά το πόσιμο νερό της βρύσης. Δεν ξέρω τώρα αν απάντησα και στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Apologies. So I think we have received a question also from... Και ο ε, Πόιτ για τις αρχές που αφορούν την μόλυνση, δηλαδή τον κίνδυνο θέσπισης αυστηρότερων παραμέτρων και το ενδεχόμενο το κόστος να τον αναλάβουν τελικοί χρήστες με βεβαίως ασφαλέστερο αλλά πολύ ακριβότερο νερό. Εδώ δεν μπορώ παρά να παραθέσω τα στοιχεία που έγιναν σε μια αξιολόγηση για την κατανάλωση και που λέει ότι η αύξηση του κόστους αν νοικοκυριό ετησίως δεν θα είναι πάνω από 7-10 ευρώ το πολύ, το πολύ. Οπότε με τη θέσπιση καλύτερης προστασίας ανθρώπινης υγείας με καλύτερες παραμετρικές αξίες δεν θα οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις όσον αφορά το κόστος για τους ε, καταναλωτές και βεβαίως πρέπει να δούμε και τα ενδεχόμενα ωφέλη και κέρδη. Γιατί όπως ξέρετε ένα λίτρο νερού βρύσης κοστίζει 0,5 cents. Και βλέπετε ποια διαφορά όταν αγοράζετε εμφιαλωμένο. Και αυτό οδηγεί σε μια εξοικονόμηση 600 εκατομμυρίων ετησίω από τα, από τα αν πίνουν ακριβώ με περισσότερη εμπιστοσύνη το νεράκι τη βρύση. Οπότε δεν βλέπω να υπάρχει κάποια προβληματική εδώ πέρα. Στο συγγνώμη αν ξέχασα τίποτα και πρόεδρε καθοδηγήστε με γιατί η εμφάνιση μου είναι παρθενική εδώ και ενδεχομένω να έχω ξεχάσει κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λέκη Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Κάνατε πολύ καλή δουλειά, κύριε Μαρό, δεν βλέπω ερωτήσει. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτές τις ερωτήσει, ε, να σα πω και το σκέλος ε, τη αναφορά των υποβολή αναφορών σε ό,τι αφορά την ποιότητα να τον υδάτων. Έχουμε την κυρία Καπεσόν Λούι και την κυρία Ρούλαντ. Η κυρία Μανφρέτη να πάρει το λόγο πρώτα να κάνει την εισαγωγή. Όντω λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο θέμα τη ε, παροχή πληροφοριών και τη υποβολή αναφορών σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υδάτων. Εδώ λάβαμε μία ερώτηση από την κυρία Καπεσόν Ρουή, Ευρωβουλευτή. η οποία ουσιαστικά ρωτά κατά πόσον έχουμε την αίσθηση ότι ενημερώνουμε τους καταναλωτές με τα σωστά εργαλεία. Ανησυχεί λοιπόν η αξία του Ευρωβουλευτή κατά πόσον βοηθάμε να μειωθεί αυτό το ψηφιακό χάσμα και όντω υπάρχει ένα άρθρο στην αναθεώρηση για την υποχρέωση που υπάρχει να ενημερώνονται οι καταναλωτέ στο διαδίκτυο. Στέκει λοιπόν ένα τμήμα του άρθρου που αναφέρεται στη σημασία για τα κράτη-μέλη να υπάρχει διαρκώς ενημερωμένη πληροφόρηση στο διαδίκτυο. Αυτό ισχύει. Αλλά υπάρχει και το άρθρο 14, το οποίο μιλάει για τη σημασία υπάρχει να ενημερώνουν διαρκώς τους ε, πελάτες τους μέσω των ε, τιμολογίων. Η τρέχουσα πρόταση λοιπόν προβλέπει τη δυνατότητα, είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Και πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό χρήζει προτέρω συζήτηση και στα πλαίσια του Συμβουλίου. Και είμαστε ανοιχτοί για να σκεφτούμε οποιαδήποτε άλλη οδό επικοινωνίας την οποία ενδεχομένω θεωρείται απαραίτητη για να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα. Ξέρετε ότι αυτό μα απασχολεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επιδιώκουμε ακριβώ στα πλαίσια τη στρατηγική για την ενιαία αγορά. Θέλουμε πραγματικά να κλείσει αυτό το χάσμα και θέλουμε όλοι οι καταναλωτέ να έχουν εμπιστοσύνη και να καταλαβαίνουν αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να κατανοούν τι ακριβώς ισχύει και να χρησιμοποιούν πιο πολύ το νερό της βρύσης. Σε ό,τι αφορά τώρα την ερώτηση της κυρίας Μπόιλαν, σε ό,τι αφορά την τάση συγκεντρώσης των ε, ζωνιακτώνων στα πόσιμα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελευταία τριετής έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε για την περίοδο 2011-2013 και η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2016. Περιμένουμε τώρα και προετοιμάζουμε την επόμενη σεφετική έκθεση, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Αυτό το καθορίζει το 13.5 του υφιστάμενου κανονισμού, της υφιστάμενης οδηγίας για τα πόσιμα είδατα. Τότε θα ξέρουμε λοιπόν πιο πολλά για την ποιότητα του πόσιμου νερού. Παρ' όλα αυτά, στη μελέτη αντικτύπου έχουμε κάποιες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Και η ανάλυση μας καταδεικνύει ότι γενικά είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό συμμόρφωσης σε όλα τα κρατημέλη σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους αναφορικά με τα ζυζανιοκτώνα, ατραζίν για παράδειγμα, και τα κτλ. Άρα ουσιαστικά σύμφωνα με τα στοιχεία του 2013 τα οποία και ανέφερα προηγουμένω, το μέσο ποσοστό συμμόρφωση σε όλα τα κρατημέλη είναι μεταξύ 99 έως 100%. Άρα και μία φορά έχουμε θετικές ειδήσει για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, λέει και Πρόεδρος για το θέμα αυτό της ε, υποβολή αναφορών. Ποιο θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Για αυτό το θέμα, κύριε Γκρουστά, θέλετε το λόγο. Ναι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι, ναι, ναι, αν μου δίνετε ένα λεπτό θα θέλω να πάρω το λόγο. Άκουσαμε την όλη συζήτηση. Και θυμήθηκα αυτό που μου πρόσφατα ένα επιστήμονα. ο οποίος εξέφρασε ανησυχίες για τα υπολείμματα ορμονών που βλέπουμε. Σε ό,τι αφορά και την επιρροή που υπάρχει στα ψάρια, σε ό,τι αφορά την επιρροή στους εφήβους, μου μίλησε επίσης και για την ε, αν θέλετε, θηλυκή διαμόρφωση, διαμόρφωση θηλυκών ε, χαρακτηριστικών στους νεαρούς άντρες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν και τοξικολογικές ε, ε, μελέτες για να δούμε πώς έχει πραγματικά το πρόβλημα, γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο είναι προφανώς κατεπήγον να το αντιμετωπίσουμε. Άλλες ρωτήσεις λέει η Πρόεδρος. Η κυρία να απαντήσει. my very expert colleagues. Οι πολλοί εμπειροί συνάδελφοι που κάθονται δίπλα μου ε, υπογραμμίζουν εκ νέου αυτά που ανέφερα και προηγουμένω, ότι με την αναθεώρηση αυτή για πρώτη φορά θα κάνουμε και θα εισαγάγουμε μια υποχρέωση ε, παρακολούθηση και κάποιων ενδοκρινικών διαταρακτών. Και επικεντρωνόμαστε στη νέα παράμετρο για τη βέτα η οποία όντω ε, θα μπορούσε να προκαλέσει τις επιτράσεις που ανέφερε η κυρία Κρουστέτε. Η νέα πρόταση λοιπόν ε, περιλαμβάνει ένα νογραμμάριο ε, αναλύτριο ως όριο. Είναι πολύ προορισμένο αυτό ως όριο. Και αυτό όχι μόνο για τις ε, ενδοκρινικές αλλά για ένα προϊόν που χρησιμοποιείται σε φαρμακευτικά προϊόντα. Παρακολουθώντας λοιπόν τη συγκεκριμένη ουσία, περιορίζουμε και την παρουσία επικίνδυνων φαρμακευτικών σκευασμάτων στην αγορά μας. Είναι μια διαδικασία εν εξελίξη. Είναι πρώτη φορά που εισαγάγεται τέτοια υποχρέωση ευρεία για παρακολούθηση τέτοιων ουσιών θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Κάθε φορά που τα κρατη που τα κρατημέλη θα συμφωνήσουν να αυξήσουν τις δραστηριότητες παρακολούθησης, θα έχουμε τη δυνατότητα να το πράξουμε αυτό. Πρόκειται για μια μεταβατική φάση την οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε, ωστόσο με κοινό στόχο της ελαχιστοποίησης του αρνητικού αντικτύπου στην υγεία των πολιτών. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Για την ε, εφαρμογή υφιστάμενης νομοθεσίας έχουμε άλλα τρία ερωτήματα. Η πρώτη. Η κυρία Σουίτσα την έφεσε για την ε, ευαισθητοποίηση για τη σπατάλη νερού. Θα θέλετε να μας απαντήσετε, κύριε Μανφρέντη. Ευχαριστώ. Όπως θα είπα ήδη, στην πρόταση αναθεώρησης δίνουμε μεγάλη σημασία στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Άρα, αφενός υπάρχει ένα άρθρο το οποίο προβλέπει στις πληροφορίες στο διαδίκτυο να συμπεριλαμβάνονται και συστάσεις και συμβουλές για την μείωση της κατανάλωσης νερού, για να υπάρξει ευαισθητοποίηση και για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η πρόταση επίσης που θα θέσαμε καλύπτει και το απόσιμο νερό, το νερό της και προβλέπει την ε, εξαρτίες σε εθνικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 13. Όπως ξέρετε, πιο γενικά σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ΙΠΑ προαγάγουν την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε υγειονομικές εγκαταστάσεις ως προτεραιότητα. Αυτό αποτελεί προφανώς και ένα από τους σημαντικότερους στόχους ε, της ε, βιώσιμης ανάπτυξης μεταξύ του 2014 και του 2020 το νερό και οι εγκαταστάσεις, ε, οι υγειονομικές εγκαταστάσεις παραμένουν κορυφαία προτεραιότητα στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, ίσως όλο μου και πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Έχουμε και πολλά περιφερειακά προγράμματα με γειτονικέ ε, χώρες ε, με την Κεντρική Ασία, με την Κεντρική Αμερική, με την Λατινική Αμερική και όλα αυτά τα προγράμματα, τα προγράμματα ανέρχονται σε αξία 800 και πλέον εκατομμυρίων. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει τη σημασία του σε ό,τι αφορά το εργαλείο αναπτυξιακή βοήθεια. Εδώ τα θέματα νερού πρέπει να πούμε ότι έχουν ενταχθεί εγκάρσια και σε άλλε πολιτικέ, γιατί υπάρχει μεγάλη σχέση μεταξύ νερού, ενέργεια, και ασφάλεια τροφίμων. Αυτά τα θέματα λοιπόν τα πραγματευόμαστε και στο πλαίσιο της ε, περιφερειακής ενοποίησης και ενσωμάτωσης, ε, μεταξύ άλλων και για το στόχο να υπάρχει ασφάλεια, σταθερότητα και περιβαλλοντική προστασία. Το Μάρτιο του 2018 ξεκίνησε μία πρωτοβουλία για να προωθηθεί στα πλαίσια της σύμβασης του ΟΕΕ η συνεργασία για το νερό. Και ο σκοπός μας είναι να υποστηριχθούν οι πεπιθήσεις μας για την κοινή αξία των διεθνών συμβάσεων σε ό,τι αφορά το νερό, δεδομένων και των αυξανόμενων εντάσσεων που επικρατούν στο θέμα του νερού. Όλοι τα ξέρουμε αυτά. Τώρα, κοιτάμε και τα κοινά ωφέλη τα οποία μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία για το νερό και από τι διεθνεί συμβάσει για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη σχετική σύμβαση του ΟΗΕ για το νερό. Και αν θέλετε να περάσω και σε μία επόμενη ερώτηση η οποία έχει κατατεθεί στο πλαίσιο αυτό, γιατί από ό,τι βλέπω έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις στην ατζέντα. Βεβαίω, βεβαίω, λέει η πρόεδρο. Δύο ε, του κυρίου Φάρια για θέματα ε, και οικονομικής ε, Ναι, ακριβώς. Ο κύριος ε, Φαρία έθεσε μία ερώτηση σε ό,τι αφορά τις ε, ακραίες που πλήττουν την Νότια Ευρώπη και σε τι επίπεδο δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντισταθμίσει τις συνέπειες των, ε, της ξηρασίας αυτές. Όπως ξέρετε, το θέμα αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερως. Έχουμε και μια ειδική ανακοίνωση την οποία δημοσιεύσαμε το 2007, το 2012. Ακολούθησε άλλη μια ανακοίνωση όπου επαναλάβαμε την δέσμευσή μας και επίσης ε, συστήσαμε και το Ευρωπαϊκό Παρτιτήριο για τις ξηρασίες. Και έτσι καταρτίζουμε καλύτερους α, δείκτες για τέτοια φαινόμενα, για τις ανομβρίες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να προαγάγει μέτρα πρακτικά για την ασφαλή και μήκο το ανακύκλωση του νερού. Θα καταθέσουμε και στην Επιτροπή σας και στο Συμβούλιο μία νομοθετική πρόταση για ελάχιστες προδιαγραφές για την ανακύκλωση του νερού και την νέου χρήση του για άντρευση. και προγραμματίζουμε να τη δημοσιεύσουμε την πρόταση αυτή το Μάιο του έτους αυτού. Σε ένα μήνα δηλαδή. Επίσης, ε, παρουσιάζουμε δυνατότητε συγχρηματοδότηση μέσω των περιφερειακών ταμείων για την αντιμετώπιση της ανομβρίας στα κράτη-μέλη. Επίση, συνεχίζουμε με τους χώρους αποθήκευσης νερού και τη χρήση πράσινων υποδομών, όπως για παράδειγμα τα φυσικά μέτρα φύλαξης νερού όπως για παράδειγμα το σύστημα φύλαξης του βρόχινου νερού. Έχουμε διάφορες έρευνες και πλωτικές μελέτες για την ε, αντιμετώπιση, για παράδειγμα, των διαρροών. Οι διαρροές αποτελούν ε, μεγάλο πρόβλημα. 23% της κατανάλωσης του νερού αποτελούν διαρροές σε όλη την Ευρώπη. Και για να σας δώσω μια συνολική εικόνα, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας σε όλη την προγραμματική περίοδο 2014 μέχρι 2020, είχαμε 670.000 ευρώ τα οποία έχουν, έχουν χρησιμοποιηθεί για διάφορα project για τη διαχείριση των υδάτων και για την ε, καλύτερη χρήση αυτών. Ελπίζουμε λοιπόν να υπάρξει ανάλογη τάση, ίσως και μεγαλύτερη τάση στο μέλλον για την καλύτερη χρήση και την καλύτερη ανακύκλωση των νερών. Και να περάσω στην τελευταία ερώτηση τώρα, μία ερώτηση που έχει να κάνει με την πρόσβαση σε ασφαλή ύδατα ως ανθρώπινο δικαίωμα. Το αίτημα η Επιτροπή να σε τους πολίτες για την πρόσβαση στο νερό αποτελεί μια σημαντική παράμετρο. Στην αναθεώρησή μας περιλαμβάνουμε μια σειρά διατάξεων που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την πρόσβαση, αλλά και με τη διαφάνεια του κόστου και των επενδύσεων που απαιτούνται για όλο το τομέα διαχείριση των υδάτων. Η αρχή την οποία και εξετάζουμε έχει να κάνει με την αρχή του να πληρώνει σε ό,τι αφορά παροχή υπηρεσιών για υδροδότηση. Αυτό προβλέπεται και στην οδηγία για το νερό, προκειμένου να υπάρχει σωστή χρέωση της χρήσης νερού στην τελική ανάλυση. Και ουσιαστικά, τι κάναμε, τι έχουμε κάνει στην αναθεωρημένη οδηγία. Έχουμε εισαγάγει κάποια άρθρα τα οποία θέλουν να δώσουν πιο πολλές πληροφορίες ε, στους πολίτες ε, για τα πόσο στα διαρροών, για το πόσο ενέργεια καταναλώνει ο κάθε πάροχος υδροδότησης, προκειμένου τελικά ο καταναλωτής να κάνει καλύτερες επιλογές. Οι διατάξεις αυτές είναι πολύ πιο φιλόδοξες ε, σε σχέση με αυτές που ισχύουν στην τρέχουσα οδηγία. Και ελπίζουμε ότι με τη σωστή προσαρμογή των διδάξεων αυτών και με τη δική σας βοήθεια θα έχουμε και θα βρούμε στο σωστό τρόπο και να ενημερώσουμε τους πολίτες, αλλά να βάλουμε και την ενημέρωση σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Μάλιστα, και τις τελευταίες δύο ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει κανείς να πάρει το λόγο. Κύριε Φαρία, Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις εξηγήσει σας, αλλά ειλικρινώς δεν είναι αρκετές. Ήμουν στο 8ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το νερό στη Βραζιλία και ήμουν ο μόνος ευρωβουλευτής παρεμπιπτόντος και όλα τα ζητήματα αυτά συζητήθηκαν εκεί και από τη δική μας την πλευρά δεν άκουσα και πολλές εύστοχες απαντήσεις. προγράμματα, ενδείξεις, μελέτες, η συνολική εικόνα από το 2014 έως το 2020, ως προς την πρώτη μου ερώτηση αυτό κυρίως, και οι άλλοι επίσης, καθώς και τα εκατομμύρια ευρώ που ξοδεύτηκαν για αυτό το αποτέλεσμα. Όμως, επί της ουσίας, τι συγκεκριμένα μέτρα έχουν αναλυφθεί Μόνο μελέτες, ακούμε, στατιστικά στοιχεία, δεν φτάνουν αυτά. Στη χώρα μου έχουμε πληγή πολύ βαριά από ξηρασίες. τα ποτάμια έχουν, ε, χάσει, έχουν στερέψει και ο κόσμος που φέρει. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας είχαμε λεψιδρία σε πόλεις. Οι πολίτες ανησυχούν Τι θα γυρίσω να πω στους πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολλές μελέτες, έχει συγκεντρώσει πολλά στατιστικά στοιχεία. Θέλουν να γνωρίζουν οι πολίτες τι θα γίνει στην πράξη για να ανακουφιστεί ε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Και το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα. Και πάλι εδώ Το θέμα είναι να μιλάμε για να, να έχουμε επίγνωση της διαρροής, των διαρροών, της πατάλης, αλλά δεν αρκεί αυτό. Και δεν απαντήσατε πάλι στην ερώτησή μου. Τι κάνατε τα χειροπιαστά συγκεκριμένα. Πολλά χρήματα μοιράζονται, ακούγονται φοβερέ ιδέε μεν, αλλά ξεκινήσαμε το 2014 και φτάνουμε στο τέλο τη θητείας. Τι συμβαίνει επί τη ουσία και συγκεκριμένα. Εάν πάτε στι νότιε χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, τα προβλήματα τα βλέπετε στην πράξη. Βλέπετε ανθρώπους χωρίς πόσιμο νερό, βλέπετε ε, ανθρώπους χωρίς πρόσβαση στο νερό λόγω έλλειψης διαφάνειας. Γιατί οι ιδιωτικές ή δημόσιες υπηρεσίες δεν προσφέρονται σε όσους δεν έχουν αρκετά για να πληρώσουν τους λογαριασμούς του. Τους κλείνουν την κάνουλα τη γενική παροχή. Μελέτες λοιπόν ωραία, στατιστικές καλά, αλλά επιτάπητος. Τι υπάρχει, αυτό θέλω να μου πείτε. Απλώς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ κυρία Μανφρέντι. δεν μπορώ παρά να δείξω ε, κατανόηση για όσα είπε ο κύριος Φαρία. Είμαι από την Ιταλία και θα ξέρετε ότι η Ρώμη, η πόλη που γεννήθηκα, ε, τον περασμένο χρόνο ήταν για λίγο καιρό χωρίς νερό. Και ο πληθυσμός προσπάθησε να αντιμετωπίσει την υπουσία νερού. Υπήρχαν προβλήματα με τις υποδομές. Καταλαβαίνω λοιπόν αυτήν την εντύπωση ανεπάρκειας που δίνουν οι απαντήσεις που έδωσα, αλλά ε, η δική μου διέστηση με οδηγεί να απαντήσω στον ε, κύριο Βουλευτή ότι θα δώσουμε λεπτομέρειες για το τι έχει ζητήσει η Πορτογαλία στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής για τα θέματα αυτά. Διότι αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολλά έχουν γίνει με πολύ συγκεκριμένα προγράμματα για να, βελτιωθεί, να βελτιωθούν οι καταστάσεις συνδροδότησης σε όλα τα κράτη-μέλη Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είστε βέβαιοι ότι όλε τι προσπάθειε που γίνονται τώρα για την ε, προετοιμασία του επόμενου πουδουπού κοιτάζει να διασφαλίσει ότι οι υποδομές υδροδότησης και το πρόβλημά τους θα αντιμετωπιστεί. Επίσης, Αυτό είναι κάτι που αφορά όχι μόνο τις χώρες του Νότου της Ευρώπης. Όταν μιλώ δημοσίως για αυτά, ε, φαίνεται να δίνεται η εντύπωση ότι υπάρχει ένα διαχωριστικό μεταξύ Βορρά και Νότου της Ευρώπης. Δεν ισχύει αυτό λειψιδρία αντιμετωπίζεται και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Ας πούμε, σε μερικές σκανδιναβικές χώρες, σε κάποιες περιοχές τους, καθώς και στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια πρόταση με ελάχιστε απαιτήσει για τη διευκόλυνση των λιμάτων, των αστικών λιμάτων που θα μπορούσαν να καθαριστούν, να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άρδευσης στη γεωργία και για άλλους σκοπούς θα θέλαμε λοιπόν να ανανεώσουμε τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης για το νερό, ένα καλό κατά την άποψή μου καταλήτη όπως θα λέγαμε για να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες δυνατές τεχνολογικές λύσεις και ε, βάσει των αρχών της κυκλικής οικονομίας να αξιοποιήσουμε όλες τις ε, διαθέσιμες πηγές νερού. Να συγκεντρώσουμε τους δυνατότερους εγκεφάλους γύρω από το ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν για τα θέματα αυτά, να συγκεντρώσουμε δηλαδή τα καλύτερα μυαλά. Θα απαντήσω πάντως στον ε, κύριο Ευρωβουλευτή ε, για τα θέματα της Πορτογαλίας με περισσότερες λεπτομέρειες και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολόκληρη, ο κύριος Βέλλα συγκεκριμένα, είμαστε πλήρως ταγμένοι στο σκοπό αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ολοκληρώσαμε το πρώτο τμήμα που αφορά την ισχύουσα νομοθεσία. Να περάσουμε τώρα στην προβλεπόμενη πρόταση οδηγίας για το νερό που προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση. Αναδιατύπωση. Η πρώτη ερώτηση αφορά την, την εγχώρια διανομή με τη σχετική αξιολόγηση κινδύνου και την έθεσε ο κύριος Βόλκεν. Και πάλι κυρία Μανφρέντι, εάν θέλετε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ερώτηση του κυρίου Βάλκεν αφορά το ζήτημα των υλικών που έρχονται σε επαφή με το νερό ως ένα μείζον θέμα, ένα μείζον πρόβλημα. Και ρωτά ποια είναι τα σχέδιά μας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό στην αναδιατύπωση. Όπως προανέφερα τα σχέδιά μας και αυτό που περιλαμβάνει η πρόταση είναι να υπάρξουν δύο παράλληλες πορείες. Θέλουμε στον αντιτυπωμένο κείμενο να διευκρινιστεί ότι η τυποποίηση, οι προσπάθειες τυποποίησης και οι τεχνικές απαιτήσεις για τα προϊόντα αυτά πρέπει να διευθετηθούν από την οδηγία για τα κατασκευαστικά υλικά και την δουλειά της τυποποίησης που γίνεται και αλλού καταλήγουμε στο πλαίσιο της ε, εκπόνησης της πρότασης αυτής ότι δεν είναι καλό για την εσωτερική αγορά να υπάρχει ε, προς το παρόν μια κατάσταση με διαφορετικές ανόμιες εθνικές πρακτικές που και μεγάλο κόστος επιφέρουν στην, ε, στον κλάδο αλλά δεν προσφέρουν ασφάλεια, βεβαιότητα, σταθερότητα στην αγορά. Δεν επιτυγχάνουμε ούτε τους στόχους της επαρκούς κάλυψης της ανθρώπινης υγείας τη ε, της ελεύθερης κυκλοφορίας των ε, εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Για το, για το λόγο αυτό εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να αναθερμάνουμε τη διαδικασία για την επιτάχυνση της διαδικασίας τυποποίησης για την υγιεινή και την ασφάλεια τέτοιων προϊόντων. Κατανοώ ότι ένα σχέδιο εντολής για τον ΣΕΝ, τον ε, Παγκόσμιο Φορέα Τυποποίησης, είναι σημαντικό μόλι, δημοσιοποιηθούν τα εναρμονισμένα, εξυγχρονισμένα πρότυπα που καταρχήν θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος της χρονιάς, θα έχουμε και μια πιο εξορθολογισμένη διαδικασία λήψη αποφάσεων για να έχουμε ασφαλή κατασκευαστικά υλικά ε, σε επαφή με το πόσιμο νερό στην αγορά να πω ότι παρά τις πιέσεις κάποιων ενδιαφερομένων και δημοσίων δεν θεω... δεν θεώρησα αρμόζων να ε, δώσουμε συγκεκριμένες περιγραφές υλικών ή τεχνολογικών λύσεων. Ακόμη χρειάζεται αρκετή δουλειά στο επίπεδο της σύνταξης της νομοθεσίας, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παραμείνει ουδέτερη ως προς την επιλογή των παραδειγμάτων και να έχει μια προσέγγιση μακροπρόθεσμη για το μέλλον. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν, βλέπει να, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλες, άλλα σχόλια για την ερώτηση αυτή. Μετά έχουμε ερώτηση της κυρίας Κάντενμπαχ. Διαδικασίες αποκατάστασης και περιορισμούς χρήσης. Θέλετε να την ε, απαντήσετε. Παρακαλώ. With pleasure, Chair. If I understand correct, actually this is a question that Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε διάφορες υποερωτήσεις στα πλαίσια αυτής της ερώτησης. Θα προσπάσω λοιπόν να τις απαντήσω όλες μαζί. Ρωτάει το μέλος του Κοινοβουλίου για το ποιες διαδικασίε παράβασης εφαρμόζονται για τις χώρες που έχουν υπερβεί τις τα όρια και τις παραμέτρους για την ανθρώπινη υγεία κτλ. Αναφέρεται η Ευρωβουλευτής στο άρθρο 3 μια νέα διάταξη της αναδιατύπωσης που καταθέσαμε η οποία στοχεύει στο να διευκρινίσει τις παραμετρικές αξίες που θα βρείτε στο παράρτημα 1 της πρότασης για να διασφαλίσουμε ακριβώς ότι οποιαδήποτε υπέρβαση αυτών των αξιών θα υποπτεύεται. Η ακριβής, διάταξη, αυτή, η ακριβής διατύπωση αυτής της διάταξης θεωρούμε ότι είναι σημαντική. Δεν λέμε ότι απλά και μόνο η υπέρβαση ε, είναι de facto απειλή, αλλά αποτελεί μια δεχόμενη απειλή στην ανθρώπινη υγεία. Οπότε οι χώρες μέλη είναι υποχρεωμένες να λάβουν δράσεις όχι μόνο με αυτά που λέει, σύμφωνα με αυτά που λέει η Υγεία, αλλά σύμφωνα και με τη βαρύτητα της κατάσταση, ενημέρωση των πολιτών, προοπτικά μέτρα άλλου κλπ. Να σας πούμε επίσης ότι γνωρίζουμε μια περίπτωση που βρίσκεται υπό διερεύνηση χώρας που αποφάσισε να διευκολύνει μια διαδικασία καθαρισμού μιας ε, ουσίας της τριαλομηθήνης και είδαμε ότι εν λόγω χώρα, σε αυτή την περίπτωση, δεν είχε επαρκώς ενημερώσει τον πληθυσμό της για την παρουσία της τριαλομεθήνης στο πόσιμο νερό. Βρίσκεται λοιπόν υπό διερεύνηση η υπόθεση αυτή και βρισκόμαστε στη δικασία παράβαση. παράβασης. Μας ρώτησαν επίσης κατά πόσο τοξικολογικά στοιχεία επιβεβαιώνουν το ότι οι παράμετροι που υπερβαίνουν σε περίπτωση που έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, αυτά αποτελούν απειλή στην ανθρωπινή υγεία. Έχουμε την τριαλομεθύνη που λέγαμε προηγουμένω. Αναγνωρίστηκαν οι βλαβερές συνέπειες αυτής της ουσίας ε, από το 1993 ήδη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Είναι μια ουσία ε, στην οποία εκτίθεται κανείς για, με διάφορους τρόπους, κατάποση, ε, η εισπνοή αέρα στους εσωτερικούς χώρους μέσω εξατμίσεις από το πόσιμο νερό, δερματολογική έκθεση, έκθεση κατά τη διάρκεια ε, ντουζ, ε, μπάνιου κλπ. Και αυτά τα υψηλά επίπεδα τριαλομεθύνης έχουν συσχετιστεί με διάφορες ασθένειες και θεωρούνται υπεύθυνα για προβλήματα υγείας, ε, σηκώτη, νεφρά, καρκίνους του στομάχου και ε, έχουν και αρνητικές ε, βλαβερές συνέπειες στα έμβρια, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Έχουμε και στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Καρκίνου που καταδεικνύουν ακριβώς τις καρκινογόνες συνέπειε αυτής της ουσίας τριγελομεθύνης. Οπότε λοιπόν μπορούμε να απαντήσουμε καταφατικά ότι πράγματι η υψηλή αξία τοξικολογικά στοιχεία και μελέτες επιβεβαιώνουν ότι αυτέ οι ουσίε οι ουσίες αυτής τη κατηγορίας αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Επίση, μα ρώτησαν οι ευρωβουλευτέ κατά πόσο θα υπάρξει μια διαδικασία μέσω της οποίας ενημερώνουν τα κρατη τους πολίτες ότι υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος και κατά πόσο μας ρωτούν αυτό θεωρείται απαραίτητο. Ήδη απάντησα όμως το ερώτημα αυτό, γιατί όπως είπα προηγουμένως ότι αυτό το άρθρο 12 αποτελεί ένα αυτόματο ε, μηχανισμό και αυτόματη κατάληξη του άρθρου του άρθρου 4 που υποχρεώνει τις χώρες ε, μέλη να θέσουν υποχρεωτικές αξίες και όρια για την προστασία της ανθρωπινής υγείας. Αλλά και πάλι είμαστε δεκτικοί να συζητήσουμε δηλαδή ακριβώς την ακριβή διατύπωση και ποιος ο μηχανισμός που θα αφορά την υπέρβαση της συγκεκριμένη αξίας του συγκεκριμένου ορίου ώστε οι χώρες αμέσως να προβαίνουν σε ενημερωτικές ενέργειες, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο. Τώρα, για το ερώτημα κατά πόσο οι διατάξεις του άρθρου 12 και η ενημέρωση του πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια των καταναλωτών, την πολλή εμπιστοσύνη στιγμές των καταναλωτών, να το συζητήσουμε κατά πόσο αυτό ισχύει ή αν ενδεχομένω ισχύει το αντίθετο. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πληθυσμού, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ενισχυμένη αφάνεια, ενισχυμένη ενημέρωση, θα πρέπει το κράτος τακτικά να ενημερώνει για θέματα που αφορούν την υγεία του γενικού πληθυσμού και πάλι όμως τονίζω ότι στην τωρινή κατάσταση ξέρετε ότι έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης και με τις υπάρχουσες παραμέτρους και νομίζω ότι παντού στην Ένωση έχουμε ψηλά επίπεδα Ποιότητα υδάτων. Και επίσης βαθμία και διαδοχικά ενισχύουμε και την αμοιβή εμπιστοσύνη με τους πολίτες ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα ενδεχομένω πανικού ή προσφυγή στο εφιαλωμένο νερό υπερβολικά. Δεν απάντησα πάντως προηγουμένως σε μια ερώτηση που αφορά τα μικροπλαστικά να σας ενημερώσω ότι μαζί με την πρόταση για την χρήση των υδάτων, αυτός είναι ένας φάκελος ε, κανονιστικός που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης εσωτερικά και μέχρι το τέλος του Μάη θα σας ε, υποβάλουμε σχετική πρόταση για τα μικροπλαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος, η κυρία Καδεμπάχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις αυτές. Καταλαβαίνω βέβαια. όπου σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους για τις επιζήμιες ε, ουσίες, ε, φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα μέτρα και άμεση απαγόρευση, αλλά αυτό δεν ήταν αυτό που ρωτούσα. Εγώ ουσιαστικά ρωτήσω το εξή. Τι θα γίνει όταν υπερβαίνονται παραμέτρους, όταν υπερβαίνονται παράμετροι ε, για χημικά ε, στοιχεία τα οποία δεν είναι επιζημία. Δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία. Εδώ βλέπω να υπάρχει μια ανασφάλεια για τέτοιες παραμέτρους στο άρθρο 12.3. Θα παραμένουν αυτές οι παράμετροι λοιπόν στο 12.3. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος μήπως για αυτό το θέμα. Όχι. Τότε κυρία Μαφρέντη παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να δώσω το λόγο στην ε, Κλεμεντίνη δίπλα μου, που το ξέρει το θέμα καλύτερα. Ευχαριστώ, λέει Κλεμεντίνη, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια παράμετρος που σχετίζεται άμεσα με την υγεία, η νοσηρότητα. και γι' αυτό ακριβώς την εντάξαμε αυτή την παράμετρο νοσηρότητας με τις υπόλοιπες παραμέτρους του παραρτήματος 1 δηλαδή στις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Πάντως ε, βέβαια θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στο πόσιμο νερό μέσω της ενημέρωσης των πολιτών σε σχέση με την υπέρβαση των παραμέτρων. Αυτό το εξετάσουμε σοβαρά. Αλλά βεβαίως και οι συνομοθέτες θα πρέπει να το δουν αυτό στις συζητήσεις στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Well, Σας ευχαριστώ. Και να περάσουμε τώρα στις υπόλοιπες ερωτήσεις για την πρόσβαση σε νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τρεις ερωτήσεις. Ρόρι Πάλμερ, Καμπεσόν Ρουίς και η κυρία Κάντιμπαχ πάλι. Κύριε Μανφρέτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή την ερώτηση, ο κύριος Πάρμερ αναφέρεται στο άρθρο 13 της πρότασης. Εκεί ορίζεται υποχρέωση για τα κρατημέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στο νερό συνολικά, αλλά προβλέπεται και δικαίωμα πρόσβασης για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν. και τι το θέμα φιλοδοξίας του άρθρου. Γενικά να σας πω ότι όλη η πρόταση έχει καταρτιστεί στα πλαίσια της επικουρικότητας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο διακριτικής ευχαίρεια των κρατών μελών στην εφαρμογή του άρθρου. Για να λάβουν ό,τι μέτρα πιστεύουν ότι είναι πιο κατάλληλα για να βελτιώσουν την εθνική κατάσταση. Έχουμε συγκεκριμένο. Έχουμε συγκεκριμένο ορισμό των εμπάρδων αυτών ομάδων, προκειμένου να τις εξυπηρετήσουμε καλύτερα. Στο άρθρο ε, 5, 8, αυτό θα πρέπει να συνάδει και με το άρθρο 18 της πρότασης και να σας πω τι λέει η πρόταση χωρίς, ε, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα των κρατών μελών να ορίσουν τις ομάδες αυτές, θα πρέπει παρόλα να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους ε, πρόσφυγες, νοματικές κοινότητες, αστεγούς, μειονότητες όπως ε, Ρώμα, Σύντη, ε, ταξιδευτές και ούτω καθεξής. Είτε έχουν μόνιμη κατοικία είτε όχι. Αυτή είναι η πρόταση που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πιστεύουμε ότι νομική, ο νομικός ορισμός στο 13.8 καλύπτει την κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε χώρα. Να σας πω πόσο ευρύ είναι το πρόβλημα το οποίο συζητάμε εδώ. Σήμερα στην Ευρώπη Έχουμε 23 εκατομμύρια κατοίκους, 5% κατά 5% των ε, πολιτών που δεν έχουν ε, άμεση σύνδεση με παροχή νερού. Μπορεί να έχουν πρόσβαση στο νερό, αλλά δεν είναι συνδεδεμένοι στο κεντρικό υδροδοτικό δίκτυο. Σε ό,τι αφορά την κατηγορία των ευαίσθητων ευαισθητοποιημένων ομάδων, έχουμε στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν ότι σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους Ρωμά έχουμε 1,6 2 εκατομμύρια άτομα σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου οργανισμού σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στο νερό. 75.000 άστεγοι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό. και περίπου 2 εκατομμύρια πρόσφυγες είναι αντιμέτωποι με το ίδιο πρόβλημα. Η πρόταση, ωστόσο, διευκρινίζει ότι είναι δικαίωμα των κρατών μελών να ορίσουν αυτές τις ευάλωτες ομάδες δεδομένης και της εθνικής κατάστασης. Να περάσω στην επόμενη ερώτηση. Στην ερώτηση της κυρίας Κάμπεσον Ρουίς. Ουσιαστικά επιστεί την προσοχή μας στο γεγονός ότι η πρόταση δεν, επεκτείνει, δεν επεκτείνεται επαρκώς ε, σε θέματα τιμολόγησης ε, του νερού και ότι δεν θα πρέπει να έχουμε δεν θα πρέπει να μελήσουμε το θέμα της ε, ένδυας του νερού. επαναλαμβάνομαι κάπως, γιατί πολλά αυτά τα θέματα αυτά είναι αλληλεσυνδεόμενα. Η μελέτη αντικτύπου για το θέμα αυτό έχει επισέλθει σε μεγάλο βαθμό λεπτομέρεια. Προσπαθούμε λοιπόν να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο σε ό,τι αφορά ε, το κόστος του νερού, σε ό,τι αφορά και το κατά πόσον είναι σωστό και αναλογικό για τις χαμηλές ή συντηματικές ομάδες. εστιαζόμαστε κυρίως στην καλύτερη ποιότητα για την ενημέρωση, γιατί το εκτιμόμενο επιπλέον κόστος ε, για κάθε νοικοκυριό είναι μεταξύ 7 και 10 ευρώ ανά νοικοκυριό. Η πρόταση λοιπόν καταδεικνύει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει θέμα υψηλών τιμών και αδυναμίας καταβολής του κόστους αυτού. Σε ό,τι αφορά την ανάκτηση του κόστους για την οδηγία για την παροχή υπηρεσιών, και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 της οδηγίας για το πλαίσιο ύδατος. Όπως ξέρετε, η οδηγία δεν προβλέπει εναρμόνιση των μέτρων για τον καθορισμό των τιμών αυτών. Παρ' όλα αυτά, σαφώς Υπάρχει η πρακτική ανταλλαγή των πρακτικών και αυτό θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε στο πλαίσιο του fitness track σε ό,τι αφορά την οδηγία, αλλά αφήνει νομίζω μια ευκαιρία για τα κρατημέλη να λάβουν υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών υδροδότησης. Για να απαντήσω λοιπόν στη συγκεκριμένη ερώτηση για το ποιου μηχανισμούς κοινωνική δράση θέλουμε να συνεχίσουμε να προωθούμε. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει συγχρηματοδότηση για τις χώρες, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν μεγάλη παρουσία περιθωριοποιημένων ομάδων, έχουμε στατιστικά στοιχεία. Ξέρουμε πού βρίσκονται αυτές οι ομάδες. Επίσης, ε, στις χώρες ε, αυτές ε, υπάρχει και η μεγαλύτερη απορρόφηση των ταμείων συνοχής στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο και φυσικά συνεχίζουμε να δραστηριοποιούμαστε με τα κρατημέλη για να υποστηρίξουμε όλα τα υποστηρικτικά μέτρα για εξασφάλιση πρόσβασης στο νερό, ιδιαίτερα για τις πιο περιτροποιημένες ομάδες. Να περάσω τώρα στην ερώτηση, αν θέλετε, της κυρίας Κάντεμπαχ. Η ερώτηση της έχει περισσότερη σχέση με τον τρόπο κατά τον οποίο η πρότασή μας απαντά στην πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών για το δικαίωμα στο νερό. Και γιατί δεν πάμε αρκετά μακριά, το μέσο της πρότασης να διασφαλίσουμε δικαίωμα πρόσβασης για όλους τους πολίτες της Ένωσης. Όντως, το άρθρο 13 κάνει λόγο για το καθήκον των κρατών μελών να βελτιώσουν την πρόσβαση για όλους και επιβάλλει και επιχρέωση διασφάλιση πρόσβαση για τις ευπαθείς και περιφερειοποιημένες ομάδες. Γιατί γιατί πιστεύουμε ότι κινούμαστε σε μία περιοχή όπου έχουμε αναγνώριση του δικαιώματος αυτού ως ενός ε, θεμελιώδης δικαιώματος όχι από τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων αλλά έχουν συμφωνηθεί τον Νοέμβριο από το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο Γκέτεμπορκ πέρσι. Είναι κάτι λοιπόν που πρέπει να γίνει για τους πολίτες και θεωρούμε ότι δεν γίνεται ένα συγκεκριμένο εργαλείο όπως οδηγία για το πόσιμο νερό να προβλέψει ένα θεμελιώδες δικαίωμα και το καθεστώς του από νομική Η οδηγία αυτή θέλει απλώς να βελτιώσει όσα ήδη υπάρχουν και νομίζω κάπως η οδηγία δίνει και πρακτικές ιδέες για λύσεις. Διότι όπως τα ξέρετε το άρθρο έχει διατυπωθεί έτσι που υποχρεώνεται τα μέλη να χαρτογραφήσουν, να αποτυπώσουν επί συγκεκριμένου χάρτη ποιε είναι οι πόλει που υπάρχουν προβλήματα πρόσβαση στην υδροδότηση και τι μέτρα πρέπει να αναλυφθούν. Θεωρούμε λοιπόν ότι ίσω επί χάρτου να μην φανήκαμε τόσο φιλόδοξοι ω προς την συγκεκριμένη διαδικασία όμω και τα μέτρα που προτείνονται και τι ιδέε που δίνουμε και την υποχρέωση που επιβάλλεται στου πολιτικού ηθήνοντε για το αν κάνουν αρκετά τα κράτη-μέλη ή όχι και τον έλεγχο που θα ασκήσουν σε αυτά είναι πολύ. Διατηρούμε ότι την προσοχή μας για το θέμα αυτό. Ελπίζω ότι απήντησα. Νομίζω ότι υπάρχει και τελευταία ερώτηση από την κυρία Πάλμερ. Άλλη ερώτηση αυτή, αλλά για αυτές τις τρεις πρώτα πρέπει να ρωτήσω εάν οι συνάδελφοι θέλουν να πούν κάτι. Κύριε Πάλμερ, ευχαριστώ δεν ξέρω αν με πείθουν αυτές οι απαντήσεις. Το άρθρο 13 είναι από τα πιο θεμελιώδη της πρότασης αυτής. Πηγαίνει στην καρδιά του αν βλέπουμε το θέμα σοβαρά. Και θέλουμε να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να ασκήσουν το θεμελιώδη δικαίωμα της κατάποσης νερού. Το άρθρο 13 προβλέπει ότι πρέπει να ε, κάνει ως υποχρέωση ένα κράτος μέλος. Αλλά μετά αυτό που προβλέπει τους επιτρέπει χειροπιαστά να μην κάνουν τίποτα. Μπορούν να εντοπιστούν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, να ενημερωθούν οι ομάδες αυτές του πληθυσμού ότι δεν έχουν πρόσβαση στο νερό, κατά πάσα πιθανότητα το γνωρίζουν ήδη, μπορεί το κράτο μέλο να αξιολογήσει τι δυνατότητε βελτίωσης τη πρόσβασης, αλλά κάνοντας το αυτό ε, από υλική σκοπιά πρακτική, τίποτα δεν αλλάζει για αυτές τις ευπαθεί, περιεθροπημένες ομάδες. Είτε είναι άστεγοι, είτε πρόσφυγες μετανάστες ή μια άστεγη μητέρα από μια ευπαθή ομάδα. Η επικουρικότητα λοιπόν εδώ είναι σημαντική και καταλαβαίνω ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν ένα ε, περιθώριο διακριτική ευχαίρεια για να εφαρμόσουν τη διατύπωσή σα, αλλά αν είναι κανεί ένα άστεγο στου δρόμου του Παρισιού ή των Βρυξελών ή του Λονδίνου και δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό ασφαλέ πόσιμο νερό, πού είναι το περιθώριο διακριτική ευχαίρεια πώς θα εφαρμοστεί σε αυτές τις ε, περιστάσεις. Με ανησυχεί λοιπόν ακόμα η διατύπωση του άρθρου αυτού, παρά είναι λόγο για το τι είναι περιθυροποιημένο και ευπαθές ε, άτομο η ομάδα του πληθυσμού. Και οι υπόλοιπε ερωτήσει το εντόπισαν επίσης. Ε, το πεδίο δράσεις που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό είναι προβληματικό. Διότι αυτό που ερμηνεύω εγώ είναι ότι όλες αυτές οι δράσεις μπορούν να εκπληρωθούν τα κατημέλη, θα έχουν συγχάσει με τι υποχρεώσεις τους, αλλά δεν θα αλλάξει καθόλου η κατάσταση για τις ευπαθεί ομάδες. Δεν αλλάζει ούτε ε, κεραία. Well, uh, Mrs. Manfredi, if you want to Κυρία Μανφρέντι, Θέλετε να απαντήσετε στο σχόλιο του κυρίου Πάλμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατανοώ, κατανοώ πλήρως. Καταλαβαίνω και τις παρατηρήσεις ε, και τα συναισθήματα και την απογοήτευση που εκφράζει ο ε, κύριος Βουλευτής. Έχω κάθε συμπάθεια για όσα λέει, αλλά διαβάζοντας το κείμενο Πιστεύω ότι έχουμε πραγματικά θέσει το θέμα ε, σωστά και σε σωστή βάση και με τρόπο σωστά εξισορροπημένο, επιτρέποντα του συνομοθέτε να γίνουν και περισσότερο φιλόδοξοι, αν θέλω και λιγότεροι, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Αλλά είμαι βεβαία ότι εάν οδηγήσετε το Συμβούλιο σε ένα φιλόδοξο αποτέλεσμα, θα το πετύχετε εσεί κυρίω. Αυτό που προτείνουμε εμεί όμω είναι αρκετά χειροπιαστό. Πρώτον, η έννοια βελτίωση πρόσβαση για όλου εντύμ, ειλικρινώς, θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, κοινοποιούν όχι μόνο το ποιες ομάδες έχουν πρόβλημα με την πρόσβαση στην υδροδότηση, αλλά και τι λόγοι υπάρχουν γι' αυτό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας πούν. Θα κάνουμε αναθεωρήσει, θα ε, υποβληθούν εκθέσει, θα γίνουν στατιστικέ όλα αυτά, συγκεκριμένα δεδομένα και μετά μπορεί να αποτελέσουν και αντικείμενο λήψη απόφαση, αξιολόγηση δυνατοτήτων για πρόσβαση στην υδροδότηση αυτών των ανθρώπων και ενημέρωσή του για τι δυνατότητε σύνδεση στο δίκτυο υδροδότηση. Συμβαίνει αυτό στα κρατη μα σήμερα. Ξέρουμε εάν τα κρατη ενημερώνουν του αστέγου πώ μπορούν να διασυνδεθούν στο δίκτυο υδροδότησης. Αυτό για το πρώτο τμήμα του άρθρου. Διαβάζω επίσης ότι ζητάμε στα κάτι μέλη να βελτιώσουν την πρόσβαση στο πόσιμο είδωρ για ανθρώπινη κατανάλωση με ενημερωτικές εκστρατείε και με δωρεάν προσφορά νερού στα δημόσια και κρατικά κτίρια. Στο συγκεκριμένο άρθρο λέει ότι τα κάτι μελη πρέπει να αναλάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να βεβαιώσουν ότι θα υπάρξει πρόσβαση για τους ευπαθείς και περιθωριοποιημένου. Στην περίπτωση που οι ομάδε αυτέ δεν έχουν πρόσβαση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει αμέσω να ενημερώσουν για την ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούν, να αναλάβουν δράση για να αποφευχθεί κάθε αντιπιθύμητη συνέπεια στην ανθρώπινη υγεία. Όλο αυτό το άρθρο που συμφωνώ μπορεί να ακούγεται κάπως ουτοπικό, καλύπτει το ίδιο θέμα με το άρθρο 16, πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Όπως ξέρετε, βάσει του άρθρου αυτού, ένα φυσικό νομικό πρόσωπο ή η ένωση, κάποια ένωση αυτών, ένωση, ενώσεις που και σήμερα κάνουν αξιέπαινη και πολύ ε, χρήσιμη δουλειά για να βοηθήσουν μειονότητες, πρόσφυγες και αστέγους, όλοι αυτοί μπορούν να προσφύγουν για να ε, διεκδικήσουν την ένωμη άσκηση των δικαιωμάτων τους αυτών. Δεν έρχομαι να πω ότι αυτό που έχουμε εδώ είναι η απίθανη καταπληκτική τέλεια λύση, αλλά έχουμε ένα πολύ σημαντικό ε, πρώτο βήμα, μπαίνουμε επιτέλους σε ένα θέμα που χρήζει της ύψης της προσοχής μας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε βέβαιοι ότι η έκβαση της νομοθετικής πρότασης θα είναι φιλόδοξη, θετική και ε, ισόρροπη, σωστά εξορροπημένη για να επιδιώξουμε την εκπλήρωση της ανάγκης που αναφέρατε. Δύο ερωτήματα έχουμε ακόμα. Μάλλον συζητήσαμε σήμερα. Άρθρο 14 Πάλμα, ενημέρωση του κοινού. Και μετά από την κυρία Κάντεμπαχ για το παράρτημα 2. Συχνότητα των ερευνών. Κύριε Μαφρέντη, Θαυμάσια θα πάτε. Ναι, προσπαθώ να τα καταφέρω όσο μπορώ, αλλά πραγματικά θα πρέπει να με ποτίσετε μετά από αυτή τη δικασία, γιατί έχω κορακιάσει. Every time I try to την ερώτηση του κυρίου Πάλμερ αυτή τη φορά που αναφέρεται στην δυνατότητα διασφάλισης καλύτερης εναρμόνισης του τρόπο με τον οποίο οι χώρες μέλη ενημερώνουν τους καταναλωτές. Αυτό που καταθέσαμε με την αναδιατύπωσή μας και εμείς αφορά νομίζω και τη βελτίωση της ενημέρωσης. Να απαντήσω λοιπόν το εξής. για την ενημέρωση online των πληροφοριών που όπως αναφέρεται μάλλον στο άρθρο 14 είναι επιλογή της χώρας μέλους. Βεβαίως εμείς δεν την προκαταλαμβάνουμε αυτή την δυνατότητα. Ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες ε, η παροχοί υδατός είναι κρατικές υπηρεσίες, έχουν δικές τους εθνικές ιστοσελίδες ε, που συνδέονται και με το Υπουργείο Υγείας της κάθε χώρας, οπότε δεν επισερχόμαστε σε αυτό το είδος, να το πω, διακυβέρνησης ή ζητημάτων διακυβέρνησης που δεν και δουλειά μας να θίξουμε. Αλλά νομίζουμε ότι υπάρχει ένα καλός βαθμός εναρμόνισης. Παρ' όλα αυτά βέβαια, όλες οι χώρες θα πρέπει να διασφαλίζουν το ότι οι πληροφορίες που ελαμβάνονται στο πράγμα 4 θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και γνωστές παντού στην Ένωση. Και όπως ξέρετε στο άρθρο 14 έχουμε προλέψει μια δυνατότητα υπό την αίρεση βεβαίω των συζητήσεων στο Συμβούλιο για την ανάπτυξη κατε... πράξεων όχι συγγνώμη, εφαρμοστικών πράξεων, εκτελεστικών πράξεων, σε σχέση με το τι περαιτέρω ή τι παραπάνω θα μπορούσε να γίνει ανάλογα με την περίπτωση. Νομίζω ότι απάντησα και στην ε, προηγούμενη ερώτηση σε σχέση με τις ε, πληροφορίες, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μόνο βεβαίως ε, διαθέσιμες online, αλλά θα πρέπει να διατίθενται και αυτές οι πληροφορίες και μέσω του λογαριασμού ίδρευσης. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις? Όχι, πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς απάντηση το ερώτημα της κυρίας Κάντεμπαχ τώρα. Ε, που αφορά κυρίως το κατά πόσο η Κομισιόν λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι έχουμε μια νέα ταξινόμηση όσον αφορά τη συχνότητα των ερευνών που έχουμε περιλάβει στην αναδιατύπωση και κατά πόσο αυτό θα οδηγήσει σε ψηλότερο κόστος για τους παρόχους ίδρευσης και ιδιαίτερα για τους μικρότερους. Να σου πω ξεκάθαρα ότι αυτή η αύξηση της συχνότητας προέρχεται από τη θαυμάσια συνεργασία που είχαμε με του συναδέλφου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για τα θέματα αυτά, οι οποίοι οι συνάδελφοι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό μα συνέστησαν να κάνουμε περισσότερα, πολύ περισσότερα. Ξέρετε ότι έχουμε τους ε, μικροβιοδείκτες που περιλαμβάνονται σε κάποιες παραμέτρους. Αλλά εδώ ακριβώς έχουμε να κάνουμε το σκέλος της αξιολόγησης. Γιατί φαίνεται ότι στους τομείς αυτούς κάνουμε λίγα πράγματα και σχετικά αργό και αργά. Μας είπε λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε το ότι γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και αυτές οι αξιολογήσεις πιο συχνά και ότι οι πάροχοι ίδρυυση θα πρέπει να κάνουν τους ελέγχους και τις αξιολογίες αυτές τουλάχιστον 10 φορές ετησίως. Και για τους πολύ μεγάλους ε, παρόχους ίδρυυσης οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να γίνονται σε ημερήσια βάση, σε σχέση δηλαδή με την αξιολόγηση της παρουσίας στο νερό βλαβερών ουσιών. Τώρα, Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Θα συζητηθεί περιττέρως πάντως το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να βρούμε μια σωστή ισορροπία μεταξύ προστασίας της ανθρώπινης υγείας αλλά και ταυτόχρονα βέβαια να αποφύγουμε την ε, δημιουργία επικαλύψεων και περί του διοικητικού φόρτου. Υπάρχει άλλο ένα ζήτημα που σχετίζεται με αυτό. Μας ρωτούν αν ξέρουμε το κατά πόσο ένας μηχανισμός ο οποίος ε, περιλαμβάνει αυτές τις τριετής ε, μελέτες για τις ουσίες, αν αυτό οδηγεί και αυτό δηλαδή σε περαιτέρω κόστος, σε αύξηση του κόστους ε, ιδιαίτερα για την παρουσία χλωρίου στο, είδα και κάποιο, στο ίδρο και κάποιων άλλων ουσιών. Ξέρουμε ότι η περίληψη αυτών των ουσιών και η εξέτασή τους σχετίζεται με την πρόταση η οποία προβλέπει θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση ανάλογα με τον κίνδυνο. Δηλαδή, θα πρέπει να διερευνούμε την παρουσία συγκεκριμένων βλαβερών ουσιών σε ε, συγκεκριμένες περιοχές μέσω δηματοληψιών. Αν λοιπόν σε συγκεκριμένες ε, περιοχές δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, τότε δεν χρειάζεται να γίνεται αυτή η υπόπτευση ανατριετία. Οπότε δηλαδή θέλουμε να είμαστε σφαιρικοί, συνολική, ολιστικοί αλλά βεβαίως λαμβάνουμε δείγματα από συγκεκριμένε περιοχές, κάνουμε προεκβολές, κάνουμε μια αξιολόγηση του κινδύνου, αλλά αν απουσιάζει από συγκεκριμένε ε, περιοχές η, η ουσία, αν δεν υπάρχει καθόλου ουσία στο νερό, τότε δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε τις αξιολογίε αυτές, τους ελέγχου αυτού Σε σχέση τώρα με το ερώτημα για το κατά πόσο Α, όχι λέει η ένα λεπτό και πάλι έχει να κάνει με το θέμα της συχνότητας. Η συμπληρωματική ερώτηση που έχω εδώ μπροστά μου αφορά και πάλι τη συχνότητα των ελέγχων των ενδατών. Εδώ μόνο θα μπορούσα να συμπληρώσω το Όπως ξέρετε, στην πρότασή μας λέμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχονται παντού και πάντα. Δηλαδή, για τις πιο επικίνδυνες ουσίες, ώστε να εφαρμόσουμε μια πολιτική μηδενικού κινδύνου. Έχουμε και το παράρτημα όμως που περιλαμβάνει και τις περιπτώσεις οι οποίες σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση. Οπότε έχουμε κάποιους υπολογισμούς που έκαναν κάποιοι και οι οποίοι μας λένε ότι θα πρέπει να, μάλλον θα αντιμετωπίσουμε αύξηση του κόστους ε, ανά πάροχο ίδρυψη γύρω στις 20.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό μας φαίνεται υπερβολικό γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη όλες οι εξοικονομήσεις που αναμένουμε από ένα σύστημα το οποίο βαθμία θα αναπτύσσεται καλύτερα και το οποίο θα είναι και καλύτερα ψηφιοποιημένο ώστε να επιταχυνθούν δηλαδή οι μηχανισμοί που αφορούν, που τους αισθητήρε. Και ταυτόχρονα συνοδεύεται αυτό από την μείωση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων τη συχνότητα υπόβολη εκθέσεων για τις χώρε μέλη. Συνολικά λοιπόν θεωρούμε ότι η πρόταση μάλλον επιφέρει μια καλή ισορροπία και δεν θεωρούμε ότι, δεν θεωρούμε ότι δημιουργεί περαιτέρω διοικητικό βάρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, νομίζω, λέει η κυρία Κάτεμπαχ θα το συζητήσουμε αργότερα, γιατί καταλαβαίνω αυτά που είπατε όμως στην ταξινόμηση των παρόχων ίδρυευσης έχουμε τους μεγάλους με 5.000 ε, πληθυσμιακή κάλυψη. Τα στοιχεία αυτά, δηλαδή τα όρια αυτά μου φαίνονται πολύ χαμηλά. Α, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ναι. Όπως λέει και η Πρόεδρος, θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Κυρία Μαρφέλτη, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και ξέρω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για σήμερα και καλή τύχη. Συνάδελφοι, τελειώσαμε με την πρωινή μας συνεδρίαση και θα τα ξαναπούμε πούμε στις 3.30 3.30 με τις ψηφοφορίες. Καλή όρεξη.